Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ορίσατε στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής μας το έτος αυτό, το 2011. Στο τέλος της συνεδρίασης είναι καλεσμένοι όλοι σε μια χριστουγεννιάτικη γιορτή στην αίθουσα και Μενούιν στις 7 το βράδυ. Η γραμματεία προετοίμασε πάρα πολύ καλό μπουφέ μην το χάσετε. Οπότε μπορούμε έτσι και εκτός συνεδρίασης να κουβεντιάσουμε λιγάκι. Ε, το σχέδιο διάταξη υπάρχει μια αλλαγή. Το σημείο 14 θα εξεταστεί αύριο. Όχι σήμερα. Έχουμε όλες τις γλώσσες εκτός από Ισπανικά, Λετωνικά και Ρουμανικά. Φτάσαμε λίγο πολύ στο ίμι τη θητεία μα και υπάρχουν αλλαγέ στην σύνθεση τη Επιτροπή μα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε ένα νέο μέλο, ένα από τα πολλά νέα, την κυρία Σοφία Μάτσε Κουκόβιτς τέος Υπουργό Υγείας της Σλοβενίας που κατά τη διάρκεια της Σλοβενικής Προεδρίας ήταν εδώ μπροστά μου. Καλώς ορίστε στην Επιτροπή μας. Έχουμε ε, μια ομάδα εργασίας για την υγεία στην Επιτροπή αυτή, όπου κυρία, ο κύριος ε, Λίζ, η κυρία Γκροστέτ και άλλοι θα χαρούν να σας έχουν μαζί τους. Χρειάζονται πάντα ενισχύσεις. Ε, από την, την ομάδα ΑΛΕ έχουμε τον Τόι Μάντας αντί της Αντίνα Μαλεάν. Και το ίδιο ισχύει για την Κρίστα Σάντελ Μόζε από την, ε, τους σοσιαλιστές που θα έρθει για να αντικαταστήσει Ροζάριο Κοντσέτα. Κατόπιν. Υπάρχει και μία αλλαγή εδώ στη γραμματεία. Βεροζέ Μποζά Είναι τμήμα της κυκλικής αναλλαγής στο σώμα και θα περάσει μια άλλη μονάδα. Θα ήθελα εδώ να πω ευχαριστώ. Βεροζέ ήταν πάντα πολύ ε, δεσμευμένη και δραστήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εργασία το τελευταίο καιρό εδώ στην Επιτροπή μας. Ναι, πράγματι, αξίζει. Französische Fernsehen will um 16.30 στις 4.30 θα έρθει εδώ η γαλλική τηλεόραση όταν συζητήσουμε τους ειδικά τροποποιημένους οργανισμούς. Δεν διαφανεί κανένα. Ωραία, θα του επιτρέψουμε να πούνε στην αίθουσα. Αύριο το απόγευμα έχουμε μία ομάδα εργασία. Τελευταία ομάδα, ε, εβδομάδα εργασία είναι, αλλά είναι μέρα εργασία. 5 με 7 για την δωρεά ιστών και κιτάρων. Καλό θα ήταν να είναι κάποιοι από εμά παρόντε είναι η έκθεση για ένα κουδάκι. Εδώ σε αυτή την αίθουσα, αύριο 3 με 5. 3 με 5. Αυτή είναι τώρα η πρώτη συνεδρίαση μετά τη διάσκεψη για το κλίμα στον Τάρμπαν. Είχαμε αποστείλει μια μεγάλη αντιπροσωπεία εκεί. Συμφωνούν όλοι. Νομίζω ότι έπαιξε πολύ καλό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήμασταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και των διαπραγματεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να ενώσει μία συμμαχία 120 χωρών. Μπορεί κανένα να τα δει τα αποτελέσματα όπως θέλει. Δεν αρκούν βέβαια για το στόχο των δύο βαθμών Κελσίου. Είναι σαφές αυτό, έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας. Αλλά δεν κατέρευσε όμως η διαδικασία, συνεχίζεται. Στην σύνοδο του Ιανουαρίου στο Στρασβούργο θέλαμε να συζητήσουμε με την κυρία Κόνι και ίσως να προετοιμάσουμε και ένα ψήφισμα. Αυτό το αποφασίσουμε οι συντονιστές αύριο το πρωί. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που θα πρέπει να προωθηθούν ακόμα και όσον αφορά την πραγματοποίηση του πρωτοκόλλου Κιώτο από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή μέχρι τον Μάιο είχαμε στον τόπο την απόφαση ότι το CCS, η ανταλλαγή αυτή θα είναι στην, ε, μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας για την καθαρή ε, ανάπτυξη. Υπήρχε μετά εκείνο το πρόβλημα για τις ε, μεταφορές εναερίως ή θαλασσίως. Για το κατά πόσο θα υπάρχει το εμπόριο των ε, δελτίων εκπομπών και γι' αυτά. Το δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, την Τετάρτη το πρωί θα αποφασίσει πάνω στην ε, προσφυγή των Αμερικανικών ε, αεροπορικών εταιρεών για το ΚΤΕΣ και τη μεγάλη συζήτηση θα πρέπει να την κάνουμε από αυτό βέβαια το Γενάρη. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών. 17 Οκτωβρίου, 26 Οκτωβρίου, 7 Νοεμβρίου και 20 22 Νοεμβρίου. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, εγκρίνεται. Περνάμε στο πρώτο πραγματικό σημείο του σημερινού απογεύματο και με μεγάλη χαρά μπορώ να χαιρετήσω την Επίτροπο για τι ναυτολικές υποθέσεις και αλία, την κυρία Δαμανάκη. Καλώς ορίσατε δεν είσαστε για πρώτη φορά εδώ, αλλά ήταν επιθυμία της Επιτροπής μας να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων μαζί σας για το θέμα της μεταρρύθμισης της Ελίας. Στο, το Σαββατοκύριακο ε, στα ΜΜΕ της χώρας μου συζητιόταν από το πρωί μέχρι το βράδυ το Συμβούλιο Αλλαγίας που μετά από 10 διαπραγματεύσεις κατάφερε να συμφωνήσει για τις αλληλευτικές ποσοστώσεις για το 2012. Αλλά η μεταρρύθμιση της ελευτικής πολιτικής συνεχίζεται βέβαια και η Επιτροπή αυτή ενδιαφέρεται για πολλούς λόγους. Βιοπικιλομορφία, προστασία των θαλασσών, προστασία των ειδών, πολλά θέματα δηλαδή ενδιαφέρουν την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, τι πρέπει ακόμη να γίνει και προς τα πού κινούμεθα. Καλώς ορίσατε λοιπόν κυρία Δαμανάκη. Θα σας δώσω αμέσως το λόγο για μια παρουσίαση και μετά θα έχουμε και χρόνο για ερωταποκρίσεις. Thank you, President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος ε, ήδη ανέφερε ότι έγιναν διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας για τις αλληλευτικές ε, δυνατότητες για το επόμενο έτος. Καταλήξαμε σε ένα συμβιβασμό μετά από δύο μερόνυχτα διαπραγματεύσεων και για να είμαι ειλικρινής, ο μόνος λόγος για τον οποίο είμαι ικανοποιημένη με αυτό το συμβιβασμό είναι το γεγονός ότι διατηρώ την ελπίδα ότι μετά από αυτή τη συμβαστική πρόταση τα κράτη-μέλη θα είναι διατεθειμένα να δεχτούν την πρότασή μας για μία εκβάθρον μεταρρύθμιση. Για να είμαι λοιπόν απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ε, σας δώσω πολλά στοιχεία προκειμένου να σας πείσω ότι οι θάλασσες και οι ωκεανοί μας ε, πραγματικά νοσούν. Όπως είπε και ο πρόεδρος ήδη, έχω ξαναέλθει στο παρελθόν και θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω και πάλι, απλώς για να καταγραφεί, ότι χρειαζόμαστε μία εκβάθρον αλλαγή διότι δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια να ζούμε με την τρέχουσα κατάσταση. Αν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, μετά από 10 χρόνια, μόνο 8 από τα 136 είδη μας θα είναι υγιή και τα παιδιά μας δεν θα μπορούν να καταναλώσουν ε, ψάρι. Και πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Έχουμε υπεραλίευση τα αποθέματά μας και η υπεραλίευση στα ευρωπαϊκά ύδατα είναι πολύ μεγαλύτερη από την υπεραλίευση σε άλλα αλλιευτικά ύδατα. Θα πρέπει λοιπόν, επειδή είμαστε υπεύθυνοι, να κάνουμε και κάτι από αυτού. Ποιο είναι το νέο στοιχείο όμως τώρα, και αυτό θα ήθελα να το επισημάνω. Από τότε που συναντηθήκαμε πέρσι, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα νέο στοιχείο στον ορίζοντα. Και το πραγματικά νέο στοιχείο είναι η οικονομική κρίση. Επομένως, Τώρα πλέον δεν τίθεται μόνο θέμα θάλασσας, δεν νοσεί μόνο η θάλασσα, νοσεί και η οικονομία μας. Και αυτό σημαίνει ότι αυτή η ριζοσπαστική αλλαγή είναι πιο δύσκολη, διότι τα πράγματα είναι πλέον πιο σύνθετα. Αυτό στο οποίο θα ήθελα να επικεντρωθώ στη σημερινή μας παρουσίαση, στη σημερινή μου παρουσίαση, είναι τα δύσκολα στάδια τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε και θα ήθελα να επικεντρωθώ κυρίως στον τρόπο με τον οποίο η κρίση επιδρά και σε εμά και στην πρόταση που κάνουμε για τη μεταρρύθμιση και τους κινδύνους που ελοχεύουν πλέον ενώπιον όλων αυτών των νέων στοιχείων και δεδομένων. Να επανέλθω λοιπόν στην πρότασή μου. Πρέπει να σας πω ότι παρά τις δυσκολίες η πρότασή μας είναι ριζοσπαστική και θα θέλαμε να παραμείνει ριζοσπαστική διότι πραγματικά χρειαζόμαστε μια νέα μεταρρύθμιση και έχω και δύο επιπλέον επιχειρήματα προκειμένου να σας πείσω ότι η νέα μας πρόταση είναι κάτι που αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε. Καταρχάς, Εάν εγκριθεί βέβαια αυτή η πρόταση, θα εφαρμόσουμε μία προσέγγιση που θα βασίζεται στο οικοσύστημα για την αλία και κατά δεύτερον θα βοηθήσουμε τον αλλιευτικό τομέα μας να ε, είναι πιο ε, βιολογικός από πλευράς ε, ε Τι σημαίνει οικοσυστημική προσέγγιση. Έχουμε τρεις βασικές δράσεις. Καταρχάς, να υπάρχει μέγιστη βιώσιμη απόδοση ε, μέχρι και το 2015 για όλα τα αλλιευτικά αποθέματα. Αυτό είναι ένας πάρα πολύ ε, βιο, ε, φιλόδοξος στόχος. Ε, να σας επενθυμίσω ότι μετά την ΑΚΟΓΙΑ ο στόχος για τη βιοπικιλότητα είναι να έχουμε μέγιστη βιώσιμη απόδοση μέχρι το 2015 οπουδήποτε αυτό είναι δυνατό εμείς έχουμε ένα πιο φιλόδοξο στόχο, να επιτύχουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση μέχρι το 2015, τελεία. Δεύτερον, θα σταματήσουν πλέον οι απορρίψεις και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, μέσο και τρίτον, υπάρχουν κάποιες διατάξεις στην πρόταση για νέο κανονισμό για κλειστές περιοχές, ε, περιοχές που θα προστατεύονται από αλίευση και αυτό φυσικά συνάδει και με την περιβαλλοντική νομοθεσία μας, διότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να συμπεριλάβουμε την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη νέα νομοθεσία. Για τα κράτη-μέλη δεν θα υπάρχει λοιπόν πλέον η ανάγκη να διατρέξουν πολλά νομοθετικά κείμενα. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι ε, μπορώ να πω ότι κινούμεθα προς μια οικοσυστημική προσέγγιση. Δεν είναι μια συνολική οικοσυστημική προσέγγιση, αλλά ε, κερδίζουμε έδαφος προς αυτή την προσέγγιση. Το δεύτερο στοιχείο που σας ανέφερα είναι ότι θα βοηθήσουμε προκειμένου να πείσουμε με πιο συγκεκριμένο τρόπο τον αλληλευτικό τομέα να ε, έχει μια πιο οικολογική, αλλιευτική πολιτική. Και αυτό ε, συμβαδίζει και με την πρότασή μας για τη χρηματοδότηση. Τον περασμένο μήνα εγκρίθηκε μια νέα πρόταση χρηματοδότησης που αφορά ένα νέο ταμείο, Ταμείο Αλληλείας και Θαλάσσιας Πολιτικής όπως το αποκαλούμε πλέον και ε, θα μπορέσουμε να έχουμε ε, αρκετά κονδύλια επαρκή θα δαπανίσουμε περίπου 6,5 δις ευρώ στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο και θα χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια αυτά με καλύτερο τρόπο ε, διότι θα εστιάσουμε και στις ανάγκες ε, της πιο οικολογικής αλληλευτικής πολιτικής. Θέλουμε να σταματήσουμε ε, το scrapping, τον παροπλισμό, να σταματήσουμε να δίνουμε κονδύλια για μεγαλύτερα σκάφη και θέλουμε να δώσουμε κονδύλια για να έχουμε μια πολιτική η οποία θα έχει μικρότερες επιπτώσεις στον αλευτικό τομέα, μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Και τι σημαίνει αυτό, καλύτερα εργαλεία, Ενισχυμένε νέες πολιτικές για αλία μικρής κλίμακας. Σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις ε, τράτες ε, στα προνόμια της χρηματοδότησης. Σημαίνει ότι μας δίνονται κάποιοι τρόποι να δράσουμε και θα διαφοροποιήσουμε και τις πηγές εισοδήματο στον αλλιευτικό τομέα. Δηλαδή θα δώσουμε στους μα μας ε, και ένα δεύτερο στήριγμα που σημαίνει ότι όταν θα κλείνουν κάποιες περιοχές αλίευσης, όταν θα κλείνουν κάποιες αλιευτικές περίοδοι για λόγους γονιμοποίησης, θα δίνουμε κίνητρα στους αλίες μας ώστε να κάνουν κάτι το οποίο έχει σχέση με την αλία και τη θάλασσα, με τα μεταποίηση για παράδειγμα των αλιευτικών ε, αποθεμάτων, ε, να υπάρχουν μηχανισμοί αποθήκευσης, ε, ε, μαγείρεμα των ε, αλευμάτων, ε, κάποια προγράμματα τουριστικά, απορρίμματα για ανακύκλωση από τη θάλασσα και θα χρηματοδοτηθούν όλες αυτές οι δυνατότητες διαφοροποίησης του εισοδήματος προκειμένου, του εισοδήματός τους προκειμένου να πιστούν ότι μπορούν να ζήσουν στη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου, ώστε να καταφέρουμε να έχουμε μέγιστη βιώσιμη απόδοση για τα αποθέματά μας. Αυτές λοιπόν είναι οι ιδέες μας και θα χρηματοδοτήσουμε αυτή τη μεταβατική περίοδο και θα πείσουμε τους αλληλείς ότι αν έχουμε μέγιστη βιώσιμη απόδοση, τότε θα έχουν και αυτοί περισσότερο εισόδημα. Και αυτό ισχύει ήδη από φέτος, ήδη συμβαίνει. Αυτό που ανέφερε ο πρόεδρος, ε, το να δώσουμε περισσότερες πισωστώσεις σε κάποιους αλληλείς, ουσιαστικά αποστέλει αυτό το θετικό μήνυμα. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικά τα είδη, ε, την έννοια των πολύ πολύτιμων ειδών. Έχουμε ήδη καταφέρει να έχουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, γι' αυτό και πλέον έχουμε τη δυνατότητα να προσδώσουμε περισσότερο εισόδημα στους αλληλείς μας. Για παράδειγμα, ε, στο Γάδο, στη δυτικά της Σκοτίας, ε, όπου καταφέραμε να αυξήσουμε τις ποσοστώσεις κατά 200% μεν, αλλά σε αντάλλαγμα θα είναι υποχρεωμένοι οι Ελλήνες να έχουν καλύτερα ε, εργαλεία. Το ίδιο ισχύει και για το γάδο στη Βαλτική θάλασσα και έχουμε και κάποια Θετικά μηνύματα λοιπόν από αυτό. Και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να αποστείλουμε. Πρέπει να πείσουμε τους πάντες ότι αν θέλουμε να κάνουμε τη μεταρρύθμιση, μετά από δύο τρία χρόνια θα καταφέρουμε να έχουμε περισσότερο εισόδημα για τους αλλήλους μας. Για την ενδιάμεση μεταβατική περίοδο ε, που θα μεσολαβήσει, θα υπάρξει χρηματοοικονομική στήριξη ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν. Αυτή λοιπόν είναι η προσέγγισή μας. Ολοκληρώνοντας, ε, θα ήθελα να τονίσω ποια είναι τα βασικά ζητήματα για τα οποία ζητάμε την υποστήριξή σας. Και το εννοώ, διότι όπως σας είπα ήδη, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η κρίση μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη μεταρρύθμισή μας. Υπάρχουν κάποια θέματα στα οποία χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας, διότι ήδη έχω την αίσθηση από τα κράτη-μέλη και από πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι όταν θα φτάσουμε στη συζήτηση στην Ολομέλεια και στην ψηφοφορία δεν θα είναι τόσο καλά τα νέα όσο θα επιθυμούσαμε. Λοιπόν, η ευάλωτη στόχη, για να το θέσω έτσι. Η μέγιστη βιώσιμη απόδοση μέχρι το 2015. Αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Τα κράτη-μέλη ήδη θα ήθελαν να υπάρχει μέγιστη βιώσιμη απόδοση μέχρι το δεν ξέρω πότε, στο διηνεκές ε, ή να εισαγάγουμε ε, κάτι το οποίο είναι πολύ χειρότερο να επιτύχουμε μεν μέγιστη βιώσιμη απόδοση, αλλά όπου είναι δυνατό, που για να είμαι ειλικρινή, σημαίνει τίποτα. Διότι τα κράτη-μέλη πάντα θα λένε ότι δεν είναι δυνατό να το κάνουν για το τάδε ή το δίνα είδος. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα χρονοδιάγραμμα για να επιτύχουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Και αυτή είναι η τελική μας θέση. Δεύτερον, χρειαζόμαστε ένα Πέρα, ένα χρονοδιάγραμμα για το βάση του οποίου θα σταματήσουν οι απορρίψει. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι επειδή λόγω της κρίσης ε, πρέπει ε, να δημιουργήσουμε ένα εθελοντικό σύστημα στις περιπτώσεις που θα ήθελε ο Αλή να συνεργαστεί μαζί μας, ναι, όλα αυτά πολύ ευπρόσδεκτα, αλλά τα δοκιμάζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν είχαμε αποτέλεσμα. Αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν είναι μια βαθμιδόν προσέγγιση, η οποία όμως θα έχει και ένα τελικό ε, χρονικό όριο και μετά στο τέλος αυτής της χρονικής περίοδου χρειάζεται απαγόρευση για τις απορρίψεις. Αυτό επιθυμούμε και γι' αυτό χρειαζόμαστε και τη στήριξή σας. Επίσης χρειαζόμαστε και πάρα πολύ την υποστήριξή σας για να μπορέσουμε να αλλάξουμε, διότι πλέον εδώ θα κάνουμε στροφή 180 μοιρών, το, η νοοτροπία που έχουμε για τα μέσα χρηματοδότησης. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσει όλο αυτό το σκεπτικό ότι δίνουμε τα χρήματα των φορολογουμένων για να κατασκευάζονται μεγαλύτερα σκάφη και να ε, χρησιμοποιούνται μεγαλύτερες ε, μηχανές, κινητήρες ε, ή πιο επιθετικά εργαλεία όπως είναι οι τράτες και ούτω καθεξής θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αλλιά μικρής κλίματα, σε ε, εξαρτήματα τα οποία ε, δεν είναι τόσο επιζήμια για το περιβάλλον και σε πιο ε, οικολογικές διαδικασίες. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας. Και ένα τελευταίο ζήτημα θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι να υπάρχει και αυτή η νοοτροπία της υποστήριξης των παράκτιων κοινοτήτων, της επιβίωσής τους της υποστήριξης της τοπικής οικονομίας στο σύνολό της και του περιβάλλοντος, προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του. Μπορεί αυτή τη στιγμή να είμαστε αντικείμενο επικρίσεων γιατί, για παράδειγμα, θέλουμε να βελτιώσουμε και να εφαρμόσουμε περιβαλλοντικά μέσα τα οποία αφορούν το Natura 2000, περιοχές απαγόρευσης αλίευσης ε, τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι αυτά είναι περιβαλλοντικά μέσα και επομένω κατά την άποψή του, η αλληλευτική πολιτική δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Εμείς πιστεύουμε το ακριβώς αντίθετο, ότι αν θέλουμε να έχουμε βιώσιμα αποθέματα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και αυτά τα εργαλεία και θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε και αυτές τις περιπτώσεις. Για παράδειγμα, θα δώσουμε μία όθηση στην υδατοκαλλιέργεια, αλλά στη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχουν και περιβαλλοντικοί κανόνες και για περιοχές οι οποίες είναι αποκλεισμένες από ξηράς, θα πρέπει να δοθούν πραγματικά μεγάλα ποσά, προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους που τίθενται από το Natura 2000 και αφορούν όλες τις ευρωπαϊκές λίμνες. Αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια σε αυτά τα ύδατα. Αυτά είναι λοιπόν ε, αυτά που έχουμε κατά νου και ελπίζω κύριε Πρόεδρε να κατανοείτε ότι χρειαζόμαστε πραγματικά τη στήριξή σας. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέδα Μανάκη για την παρουσίαση αυτή τη τόσο σημαντική αυτή μεταρρύθμιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη-μέλη ήταν στην Αγκόγια, όπου υπήρχε μια επιτυχής ε, ολοκλήρωση μια διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών και η Ευρώπη ανέλαβε την υποχρέωση να αναπτύξει την ε, βιοπικιλομορφία, ιδίω να προστατεύσει την βιοπικιλομορφία στην θάλασσα, με προστατευμένες περιοχές και με άλλα μέτρα. Λοιπόν, υπάρχουν πολύ καλά επιχειρήματα. Αναφέρατε τα, τα κύρια σημεία, σίγουρα θα επανέλθω σε αυτά οι συνάδελφοι. Θα περάσουμε λοιπόν τώρα στους ομιλητές που έχουν το λόγο. Καταρχήν, η κυρία Φωνσβάς Γκοστέτ. Καλημέρα σας. Δύο λεπτά ο καθένας. Αλλιώς δεν θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε που ήρθατε εδώ μεταξύ μας για να ανταλλάξουμε απόψεις για ένα θέμα πάρα πολύ λεπτό και ευαίσθητο, την αλληλεία για χώρες ε, που έχουν θαλάσσιες ακτές τουλάχιστον. Συμφωνούμε πλήρως με τις μεγάλες αρχές τις οποίες απαριθμίσατε την οικοσυστημική προσέγγιση, τον προσανατολισμό προς μια πιο οικολογική πολιτική, αλλά έχω μερικές ανησυχίες σχετικά με τις παραχωρήσεις, τις αλλιευτικές που μεταβιβάζονται, τις μεταβιβάσιμες, διότι διαρωτώ με αν αυτό θα έχει αντίθεση αντίκτυπο πάνω στις ποσότητες που αλλιεύονται, διότι φοβούμε ότι οι ποσοστώσεις, εφόσον θα υπάρχει ένα σύστημα ποσοστώσεων, αν κατάλαβα καλά, οι ποσοστώσεις θα συγκεντρωθούν στα χέρια των μεγαλύτερων εφοπλιστών που και, που, κινδυνεύουν οι μικρές αλλιευτικές επιχειρήσεις, μπορεί να τις αγοράσουν. Είπατε στο τέλος ότι θα θέλατε εμείς να σας υποστηρίξουμε για την βιοτεχνική αλληλεία, συμφωνούμε, διότι αυτή παίζει οικονομικό και κοινωνικό ρόλο στα μικρά αλλιευτικά λιμάνια και πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Έχω λοιπόν αυτή την ανησυχία σχετικά με την βιώσιμη μέγιστη απόδοση, είναι ρεαλιστικός στόχος, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση κατά αλληλεία, ε, διότι για να λάβουμε υπόψη τις συστάσεις των διασκέψεων της Ναγκόγια και του Johannesburg σε σχέση με τις απορρίψεις, ε, ο στόχος μου φαίνεται πάρα πολύ καλός, θα πρέπει ε, να περιορίσουμε τις απορρίψεις στη θάλασσα, αλλά τα σκάφη, κυρίως αυτά της βιοτεχνικής αλίας, είναι εξοπλισμένα για να μπορέσουν να κρατήσουν αυτά που θα πρέπει να απορριφθούν. Νομίζω ότι εκεί θα υπάρξουν προβλήματα. Ήθελα λοιπόν να σας προειδοποιήσω για το θέμα αυτό. Πολύ ωραία, πολύ καλή ερώτηση. Ο Κρήτον έχει το λόγο. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Επίτροπο. Χωρίς καμιά αμφιβολία τα όσα είπατε, είναι σημαντικά. Ε, δεν πρέπει να υπάρξει μια εκβάθρον ε, μεταρρύθμιση για να μην μειωθούν τα αποθέματα και υπέρ των ε, παράκτιων κοινοτήτων και για όλους μας. Εν μια από τις ιδέες που έχει περισχύσει στην Επιτροπή Αλίας είναι η ιδέα των αλλιευτικών αποθεμάτων δηλαδή περιοχές κλειστές όπου θα υπάρχουν απαγορεύσεις αλίας, όπου θα μπορούν να αναπαραχθούν ε, τα ψάρια και θα μπορούν να μετακινηθούν ευκολότερα ε, σε αυτή την περιοχή, διότι υπάρχει αυτή η αναπαραγωγή, η αναγέννηση, γεμίζει ο άδειος χώρος. Νομίζω ότι αυτό, αυτό το σύστημα θα είναι καλό να εφαρμοστεί ως υποχρέωση διότι υπάρχει κατά το μάλλον ήτον στην πρόταση ως εθελοντικό εργαλείο, αλλά θέλουμε να, είναι, ε, κάτι, να είναι κάτι το υποχρεωτικό για τα αλλιευτικά αποθέματα. Ποια είναι η θέση της Κομισιόν ε, όταν θα έρθει μια τέτοια πρόταση από το Κοινοβούλιο για τις διαπραγματεύσεις. Chris Davis ε, για τα fish and chips. Ευχαριστώ κύριε ε, Πρόεδρε. Θα αφήσουμε τα chips, ε, τις πατάτες κατά μέρος, θα ασχοληθούμε μόνο με τα ψάρια. πριν από μερικές μέρες η Επιτροπή είχε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και είχαμε κοινικότητα στην στάση ορισμένων κρατών μελών σε σχέση με την αηφόρο βιώσιμη ανάπτυξη και μεταρρύθμιση και είναι δύσκολο να εξαλειφθούν ορισμένες αντιρρήσεις. Βεβαίως υπάρχει υποστήριξη αυτής της Επιτροπής και χάρηκα ε, με τις απόψεις της Φρανσουάς Γκροστέτ και την υποστήριξη που σας έδωσε ως εκπρόσωπος της Γαλλίας. Δύο θέματα κυρίως θα ήθελα να επισημάνω ε, μέχρι το 2015 ο στόχος είναι πάρα πολύ καλός, αλλά θα ήθελα να πάω πέραν αυτού. Ε, δεν θέλουμε να ε, γεμίσουμε και πάλι τις θάλασσες με ψάρια, να πηδάνε τα ψάρια πάνω από τη θάλασσα ε, για να έχουμε λιγότερες εισαγωγές αλλιευτικών προϊόντων. Θα ήθελα να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Γιατί πήγατε πέραν του MSY για, σε σχέση με αυτήν την φιλοδοξία. Ε, χρειάζεστε ε, σχέδια μακροπρόθεσμα διαχείρισης. Είπατε αλλού ότι η Επιτροπή δεν θα είναι σε θέση να έχει τέτοια σχέδια μακροπρόθεσμα για όλους τους τομείς της Αλληλίας μέχρι το 2020, το 2018. Ε, δεν θέλετε ίσως την αρχή της προφύλαξης εντωμεταξύ. Τι κάνουμε πώς ε, θα έχετε ε, NSY μέχρι το 2015 όταν δεν έχουμε αυτά ε, τα σχέδια, πώς θα έχουμε την μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Όσον αφορά ε, τις ανταλλαγές ε, των δικαιωμάτων. Το non-paper λέει ότι αφού ε, λήξει ο χρόνος θα επανέλθουν τα ποσοστά αυτά στις χώρες μέλη. Μίλησα και με τους Σουηδούς. Όλοι έχουν TFC με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Πώς θα, τι θα κάνετε για να εξασφαλίσετε ότι μια εταιρεία, ας πούμε, η οποία έχει μια παραχώρηση αλλιευτική, ε, τι θα κάνει, θέλει να εξασφαλίσει ότι θα υπάρξουν στο δυνατόν ε, περισσότερη ποσότητα, περισσότερα αποθέματα. Τι θα γίνει μετά από 15 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Γιώζε Μανουέλ Φερνάντες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ την ε, κυρία Επίτροπο και την ευχαριστώ που βρέθηκε μεταξύ μας σήμερα το απόγευμα. Θα ήθελα να μου πείτε εάν στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές θα υπάρξει κάποια σύνδεση με την πολιτική συνοχή για την αλία μικρής κλίμακας, διότι υπάρχουν επενδύσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές, παραδείγματος χάρη για την μείωση της λάσπης και θα ήθελα να υπάρχει περισσότερη ε, διασύνδεση ανάμεσα στην αλλιευτική πολιτική και την πολιτική ε, συνοχή. Οι μικρές επενδύσεις στις ακτές είναι πάρα πολύ σημαντικές όχι μόνο ούτω ώστε να υπάρξει δυνατότητα αλλίας, αλλά επίσης για να μπορέσουμε ε, να επιτύχουμε τους στόχους της στρατηγικής 2020 για τις θέσεις εργασίας, για την κοινωνική συνοχή και επίσης για τον τουρισμό. Ήθελα επίσης να ρωτήσω σε σχέση με την αλληλεία μικρής κλίμακος, τι νέα μέτρα θα είναι διαθέσιμα στις ε, δημοσιονομικές προοπτικές ε, σε ποσοτικά μεγέθη. Θα, πρέπει να θα ήθελα να περάσω και σε ένα δεύτερο θέμα. Ε, νομίζω ότι σε σχετικά με την συμφωνία αλίας με το Μαρόκο, η παράταση που δέχθηκε και το Κοινοβούλιο, κακώς νομίζω, τι σκέφτεται η Κομισιόν να κάνει. Και αν πιστεύει ότι αν θα έπρεπε οι αποβάσεις αυτές, οι φορτώσεις, εκφορτώσεις θα έπρεπε ε, να επιτρέπονται και ε, τι σκέφτεται η Κομισιόν για να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Bill Newton Πριν από μερικά χρόνια πέρασα μια εβδομάδα σε μια τράτα στην Βόρειο Θάλασσα. Ίσως δεν είναι αφελής η ερώτηση, αλλά μερικά από τα αλλιεύματα ε, πρέπει να απορριφθούν δεν θέλουμε να εκφορτωθούν ορισμένα πράγματα, ορισμένα προϊόντα τα οποία δεν χρειάζονται. Τι ε, προτείνεται σχετικά με την θέση σε εφαρμογή. Η θέση σε εφαρμογή, η επιβολή των μέτρων επαφίεται στα κράτη-μέλη αλλά τι ε, βεβαιότητα μπορούμε να έχουμε ότι τα κράτη-μέλη θα κάνουν αυτό που έχουν υποσχεθεί να κάνουν, που υποχρεούνται να κάνουν βάσει ε, της νομοθεσίας. Υπάρχουν κυρώσεις, υπάρχει κάποια τιμωρία σε σχέση με τις ε, ποτοστώσεις, υπάρχει κάποια επιθεώρηση, διότι είδα το σύστημα δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Ευχαριστώ πολύ. Εντίτε Στρέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Επίτροπο και να την συγχαρώ για τις προσπάθειες ούτως ώστε να συμφιλειωθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι με τα νόμιμα συμφέροντα των αλλιέων. Και με βάση αυτές τις αρχές θα ήθελα να τη ζητήσω να διευκρινίσει λίγο περισσότερο τι εννοεί ε, με απόδοση ε, βιώσιμη και με την υδατοκαλλιέργεια. Αυτό το οποίο θέλουμε να επιτύχουμε είναι περισσότερες, ε, περισσότεροι αλλιευτικοί χώροι, περισσότερη υδατοκαλλιέργεια, αλλά χρειάζεται περισσότερη σκέψη, περισσότερα μέτρα. Η αηφορία από περιβαλλοντική απόψεως είναι κάτι που έχει αμφισβητηθεί και έχω ένα άλλο ερώτημα που έχει σχέση με την αλία μικρής Ε, Έγινε λόγος από την Επιτροπή για στήριξη σχετικά με τις εκφορτώσεις. Διερωτώ με, την αλία μικρής κλίμακος αν δεν θα υπάρχει πλέον καμία οικονομική υποστήριξη ε, για τον εξυγχρονισμό των σκαφών, διότι είναι νομίζω η, η μικρή μικρής κλίμακος είναι η πιο ευάλωτη και αν δεν λάβουν κάποια στήριξη από κοινοτική θα βρεθούν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση σε σχέση με την αλληλεία μεγάλη κλίμακας. Ευχαριστώ. Αυτό που θα είναι δύσκολο είναι ότι όλοι θα πούνε ότι θέλουν να εφαρμόσουν την κοινή ε, αληφτική πολιτική, όλοι θέλουν, ε, θα πούνε αληφορία, αλλά στις λεπτομέρειες δεν θα είναι κανένας υπέρ. Πόσο η φόρο ήταν το Συμβούλιο αλληλιά την περασμένη εβδομάδα κατά τη γνώμη σας. Εσείς ε, ποια άποψη έχετε για την αηφορία των αληφτικών ποσοστώσεων που αποφασίστηκε την περασμένη εβδομάδα. Μετά, πολλοί λένε ότι πρέπει να κάνουμε τα πράγματα κάπως διαφορετικά, θα πρέπει να είναι ανηφόρα. Είναι άνοιχτη η Κομισιόν για άλλου είδους προγράμματα, μεταφορά των δικαιωμάτων κλπ. Αν κάποιος δηλαδή πει, έχουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο, επίσης αηφόρο όμως, επίσης βιώσιμο. Θα το υποστηρίξετε, θα το εξετάσετε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα κάποιος από μια μεγάλη αλληλευτική χώρα. Ο Ρίχαρτ Ζέμερ από την Αυστρία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για το καλό βαθμό. Αλλά και σε εμά τρώμε πολύ ψάρι και θέλουν και οι δικές μας χώρες να μπορούν να έχουν ψάρι στο πιάτο τους. Η ερώτησή μου, κύριε Επίτροπε, έχει το εξή. Τήρεται πάντα το θέμα της βάσης δεδομένων. Ακούσαμε διάφορα στη συζήτηση. Κατά την γνώμη αρκεί ένα έτος το 2015 για όλα τα είδη να έχουμε εκεί την μέγιστη απόδοση οικονομικά. που θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε αναείδος. Δεύτερον, η εφαρμογή. Άμα δω τι γίνεται με την Ισλανδία, παραδείγματος χάρη. Πέτυχε την βιωσιμότητα αυτή. Τι θα μπορούμε να κάνουμε εμείς όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα ριζοσπαστικό μέτρο. Πώς θα το εφαρμόσουμε όμως πραγματικά. Και κατά πόσον τώρα αυτή η μικρή βιοτεχνική αλία είναι η πραγματική λύση, δεν ξέρω. γιατί θα πρέπει οι αλληλείς να μπορέσουν να επιβιώσουν οικονομικά. Αυτό εξαρτάται από κάθε περιοχή. Δεν θα ήταν λοιπόν ο κύριος στόχος του Συρικού Ταμείου να προωθήσει τον σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί νομίζω τα μικρά λεφτικά σκάφη δεν θα έχουν δυνατότητες επιβίωσης μακροπρόθεσμα. Σας ευχαριστώ. Πέστε. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν όσον αφορά την ανευτική στη συμφωνία με το Μαρόκο. Σπάνια χάρηκα στη ζωή μου τόσο όσο την περασμένη εβδομάδα. Γιατί καταφέραμε κάτι πολύ σημαντικό, την παράταση δηλαδή. Αυτή η συμφωνία είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρώ ότι η Κομισιόν θα σεβαστεί την απόφαση του Κοινοβουλίου και δεν θα υποβάλει τίποτα το καινούριο. Η Κομισιόν θα πρέπει να φροντίσει να τηρούνται οι διεθνείς συμφωνίες. Έχει κάθε συμφέρον γι' αυτό. Τώρα, όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της Ελίας, ορισμένοι συνάδελφοι ανέφεραν σημαντικά σημεία και εγώ θα ήθελα να τονίσω ένα από αυτά το θέμα της δυνατότητας εποπτείας μπορούμε να συστήσουμε διαμακρών και να ορίσουμε στόχους, αλλά θα πρέπει να έχουμε μια πραγματική δομή τελικά, μια δομή η οποία θα μας επιτρέψει να ελέγχουμε τα ύδατα. και τη σχετική τροποποίηση της εργασίας μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω. Πρέπει να υπάρχει ο σωστός ε, έλεγχος και εποπτεία, ώστε τα κράτη-μέλη να μην εφευρίσκουν συνεχώς κανόνες για να μην χρειαστεί να τηρήσουν τη μία την άλλη διάταξη. Τώρα, ρευτικές ποσοστώσεις. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με αυτά που ελέγχθησαν. Υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι οι μεγάλες εταιρείες να εκμεταλλευτούν αυτές τις ποσοστώσεις. Εμείς θέλουμε όμως να ε, υποστηρίξουμε την βιοτεχνική αλληλεία και είναι περίεργο να μπορεί κανένας να αγοράζει αυτά τα, αυτά τα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ο Καρλ Σλούτερ. Θα σας καλωσορίζω εδώ και θα ήθελα να επαναλάβω τα που ακούστηκαν για τη Δυτική Σαχάρα. Και επίσης αναφερθήκατε σε μια προσέγγιση ανά οικοσύστημα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση αυτή. Αυτό σημαίνει όμως, εδώ είμαι, στο πλάι. Αυτό σημαίνει, λέω, ότι θα πρέπει να τονίζεται και το θέμα της χημικής μόλυνσης που διαταράσσουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Λοιπόν, θα ήταν καλό να μας βοηθήσετε να προστατεύσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον γιατί αυτό σχετίζεται βέβαια με το θέμα της Ελίας. Κατόπιν, το θέμα των αυτοφορολογικό. Ε, Αυξήθηκε η φορολογία στο 79% των περιφερειών και ειδών. Ξέρουμε όμως ότι Ε, το θέμα, ε, συγγνώμη, το θέμα δεν είναι το φορολογικό, το θέμα είναι οι μέγιστε ε, αλευόμενες ε, Δεν ξέρω γιατί αυξάνονται, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει υπεραλλήλεια. Θα ήταν καλό να έχετε στον κάθε έναν, στον κάθε ένα πολίτη να δώσετε μια τέτοια ποσόστοση και αν κάποιος θέλει να είναι επαγγελματίας ελαιάς θα πρέπει να έρθει σε εμά όλους που ο καθένας έχει αυτό το, το τάκ, αυτή την ποσόσταση και να αγοράσει την ποσόστοση. Αυτό θα ήταν πιο λογική προσέγγιση. Είδα το καλλιέργειες. Ε, την περσμένη θητεία είχα κάνει μια σχετική έκθεση. Αν θέλουμε δηλαδή να απαγορεύσουμε τις, ε, τις απορρίψεις, θα πρέπει να δούμε το θέμα της υδατοκαλλιέργειας, να τα συσχετίσουμε τα δύο αυτά. Sorry. And if I have to leave before you... Και με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εάν, εάν αναγκαστώ να φύγω πριν απαντήσετε, απαντήστε μου και ε, ο βοηθός μου να το γράψει. Σίγουρα, σίγουρα θα τη γράψουμε την ε, απάντηση. Άννα Ρόσπαχ, πρώτη τελευταία μιλήτρια. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποβάλω μία σύντομη ερώτηση. Έχετε γνώση, στατιστική στοιχεία ή οτιδήποτε κατά πόσον γίνεται εμπόριο των ποσοστώσεων στον ίδιο τρόπο στο βορρά της Ευρώπης όπως και στο νότο της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Και τελευταίο, ο Τζιμ Νίκερσον, αλλιέας από την Βόρεια Ελλαδία. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι έχει δίκιο ο Επίτροπος που τονίζει ότι είναι ε, πολύ άσκημη εποχή τώρα με την οικονομική κρίση. Μπορούμε βέβαια να κάνουμε πολλά πράγματα πολύ καλύτερα από το κάνουμε στο παρελθόν. Υπάρχουν πάντα έντονες διαφωνίες μεταξύ των αλλιών και των επιστημόνων. Αυτό είναι επιχείρημα που ακούγεται εδώ και χρόνια πριν έρθετε εσείς εδώ και γίνετε επίτροπος. Χρειαζόμαστε βέβαια για τη μεταρρυθμίση καλύτερα επιστημονικά στοιχεία. Ε, στην Ολλανδία έχουμε στοιχεία επιστημονικά και μου λένε ότι τελικά ήταν ανεύθυνα τα στοιχεία αυτά. Δεν χρειαζόταν να τα ακούει κανένας γιατί υπήρχαν κάποια βλέμματα στις Ιλλανδικές θάλασσες λόγω των επιστημονικών στοιχείων. Τώρα είχε κλείσει η Ιρλανδική θάλασσα 7 χρόνια και δεν έχουμε επανέλθει στα κανονικά στοιχεία, στα σωστά στοιχεία, στις σωστές ποσοστώσεις. Μπορείτε να μου πείτε κάτι πάνω σε αυτό. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω την απάντησή σας. Είναι εύκολο βέβαια να είμαστε εδώ στις Βρυξέλλες και να συζητάμε για τα πάντα. Αλλά αναρωτιέμαι, γιατί θα πρέπει οι, οι αλληλείς της Ευρώπης να έρχονται εδώ στις Βρυξέλλες ε, πρώτη και δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου για να ακούσουν κάποιες λύσεις. Οι μικρές κοινότητες εξαρτώνται από αυτά και εκεί που προέρχομαι εγώ, οι μικρέ κοινότητε αυτέ δεν έχουν καμία εναλλακτική λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επίτροπε, πολλέ ερωτήσει έχετε. Πολύ υποστήριξη όπω είδατε. Παρακαλώ στι απαντήσει σα. Ωραία. Να περάσουμε κατευθείαν στο ψητό, να μην χάσουμε χρόνο. Καταρχά, τα μεταβιβάσιμα δικαιώματα. Να σα δώσω κάποιε πληροφορίε και κάποιε εξηγήσει. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε μέσω αυτού του συστήματο είναι να προτείνουμε στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να μπορούν να μεταβιβάσουν δικαιώματα βάσει κάποιων αρχών οι οποίε θα ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη θα εισαγάγουν το σύστημα και θα έχουν την ευελιξία να το κάνουν με τον τρόπο τους μεν, αλλά υπάρχουν κάποιες αρχές οι οποίες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα πρέπει να υπακούονται. Και αυτό είναι αυτό το οποίο είχαμε απαντήσει ακριβώς, κύριε Σλίτερ, αν ε, λέω σωστά τον επιθετό σας. Εμείς θεωρούμε ότι η αλία είναι δημόσιο αγαθό. Τα αλλιευτικά αποθέματα αποτελούν δημόσιο αγαθό. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει αυτά τα δικαιώματα στους πλειοκτήτες για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποφασίσουν και από εκεί και πέρα μπορούν να τα ε, άρουν εάν ο χρήστης των δικαιωμάτων δεν, χρησιμο... Ε, δεν συμπεριφέρεται σωστά, δεν τα χρησιμοποιεί καταλήλως. Αυτό είναι το σκεπτικό. Δεν θα παραχωρήσουμε στους πλειοκτήτες ένα δικαίωμα ιδιοκτησίας θα τους δώσουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα δημόσια αποθέματα, διότι τα αλλιεύματα είναι δημόσιο αγαθό. Δεν ε, υπάρχουν ομοιότητες εδώ με τη γεωργία ή με άλλους ε, τομείς, διότι στη γεωργία καλλιεργούμε ε, σπόρους ή οτιδήποτε άλλο, φρούτα, εκεί είναι κάτι το οποίο υπάρχει. Είναι μια δημόσια πηγή και θα τους δώσουμε το δικαίωμα να τη χρησιμοποιούν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εάν συμπεριφερθούν σωστά, θα έχουν αυτό το δικαίωμα για περισσότερο χρονικό διάστημα. Εάν δεν συμπεριφέρονται όπως πρέπει, τότε θα τους αφαιρέσουμε τα δικαιώματα. Για να απαντήσω λοιπόν και στην ερώτησή σας, ε, το σκεπτικό μας δεν είναι ότι θα τους ε, ε, αφαιρέσουμε όλα τα δικαιώματα μετά από ένα χρονικό διάστημα, αλλά θα αφαιρεθούν τα δικαιώματα εάν οι πλειοκτήτες δεν έχουν τηρήσει τους κανόνες. Είναι ένα μέτρο συμμόρφωσης με τον ένα με τον άλλο τρόπο και βάσει των αρχών μας θα υπάρχουν και κάποιες ρήτρες ασφαλείες για να μην υπάρχει ε, συγκεντρωτισμός των δικαιωμάτων για να απαντήσω και σε μια άλλη ερώτηση από την κυρία Γκροστέτ. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν είναι να τους δώσουμε το δικαίωμα να αλλιεύουν, αλλά ταυτόχρονα θα υπάρχουν και δικλείδες ασφαλείας. Για παράδειγμα, μπορεί να εξαιρείται η μικρή κρίμακα ασφαλεία από το σύστημα ε, παντελώς, να μην υπάρχει θέμα δικαιωμάτων εκεί. Ή η μικρή κλίμακα ασφαλείας θα μπορεί να κάνει εμπορία δικαιωμάτων μόνο μεταξύ άλλων αλλιών μικρή κλίμακα. Ή ε, οι πλειοκτήτες να μπορούν να έχουν μόνο δύο ή τρία δικαιώματα, επί παραδείγματα. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας λοιπόν κατά του συγκεντρωτισμού και ε, υπέρ τη προστασία τη μικρή κλίμακα ηλία. Υπάρχουν δικλείδε ασφαλείας ώστε τα λευτικά αποθέματα να είναι δημόσια ιδιοκτησία. Αυτή είναι η πρόθεσή μα. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές παρανοήσεις εδώ και ε, δεν είστε και κατάλληλα ενημερωμένοι νομίζω. Αλλά πρέπει να συνεργαστούμε ώστε να εξεύρουμε την καλύτερη λύση. Ε, για να είμαι ειλικρινή, το θέμα είναι ιδιαίτερα διαφιλονικούμενο και ε, αν υπάρχουν κάποιες θετικές προτάσεις ε, είμαι στη διάθεσή σας να προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για τις απορρίψεις τώρα. Χρειάζεται ένα τελικό χρονικό περιθώριο. Τι σημαίνει αυτό ότι όταν θα σταματήσουν οι απορρίψεις, οι πλειοκτήτες θα πρέπει να εκφορτώνουν τα πάντα, να εκφορτώνουν ό,τι αλλιεύουν. Και τι σημαίνει από εκεί και πέρα. Εάν αυτά τα οποία εκφορτώνουν, ή μάλλον πρώτον, θα τους δώσουμε ε, επιδότηση, πολύ γενναιόνορη, για να υπάρχουν ε, χώροι αποθήκευσης. Και εκεί μπορεί να αποθηκεύουν ό,τι αλλιεύουν. Ό,τι μπορεί να απολυθεί, απολύτε αλλά για παράδειγμα μπορεί να εκφορτώσουν και γόνο. Και εμείς δεν θέλουμε να πωλείται γόνος διότι θα δημιουργηθεί αγορά για γόνο. Αυτό λοιπόν που θέλουμε είναι να τους δώσουμε τη δυνατότητα να τα συγκεντρώνουν κάπου και να τα χρησιμοποιούν ως ε, ε ηχθιάλευρο να μην μπορούν να το πουλήσουν. Τι άλλο θα κάνουμε, θα τους δοθεί η δυνατότητα να συγκεντρώνονται όλα αυτά κάπου και από εκεί και πέρα να ε, χρησιμοποιούνται για νέες τεχνολογίες. Για παράδειγμα υπάρχει τώρα αυξανόμενη ζήτηση για λιεύματα για την παραγωγή κολαφώνου ή και άλλων ε, υλικών, ουσιών σε φαρμακευτικές βιομηχανίες. Μπορούμε να βρούμε λοιπόν εναλλακτικέ λύσεις. Το σκεπτικό μα είναι όμω ότι θα εκφορτώνονται τα πάντα και αυτό θα είναι όταν θα εκπνεύσει η προθεσμία, το χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει. Στο τέλο αυτού του χρονοδιαγράμματο όσοι πλειοκτήτε θα είναι υποχρεωμένοι να εκφορτώνουν τα πάντα. Όσον αφορά του τρόπου ε, δημιουργία και εισαγωγή αυτών των ε, fish reserves, των καταφυγίων για τα αλλιεύματα. Θα προσπαθήσουμε ναι, να δημιουργήσουμε τέτοιους χώρους, αλλά υπάρχουν κάποια νομικά προβλήματα τι θα κάνουμε. Θα δώσουμε στα κράτη-μέλη, διότι αυτό δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, είναι αρμοδιότητα του κράτους μέλους, θα τους δώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα να αποφασίσουν από αυτόν σε περιφερειακό επίπεδο. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, όλα τα κράτη-μέλη γύρω από τη Μεσόγειο θα μπορούν να αποφασίσουν από κοινού και αν συμφωνήσουν να υπάρχουν αυτές οι κλειστές περιοχές απαγόρευσης αλίευσης, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίσει να τα δεχτεί. Αυτό είναι απάντηση και στις παρατηρήσεις που άκουσα ότι πρέπει να έρθουν όλοι οι αλληλεί εδώ στις Βρυξέλλες και να αποφασίσουν όλα εδώ στι Βρυξέλλες τέρμα αυτό. Δεν χρειάζεται να έρχονται όλοι στις Βρυξέλλες. Ε, θα μπορούν να αποφασίζουν σε περιφερειακό επίπεδο και εμείς θα υποχρεούμε να τηρήσουμε αυτές τις συμφωνίες αν υπάρχουν. Εάν δεν υπάρχουν όμως συμφωνίες ε, για κλειστούς χώρους ε, όπου θα απαγορεύεται η αλίευση, τότε εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Προσπαθούμε να βρούμε ε, μία νομική διέξοδο για να μπορούμε να παρεύουμε στις περιπτώσεις που τα κράτη-μέλη διστάζουν να αποφασίσουν ε, για αυτές τις προστατευόμενες περιοχές. Για τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση τώρα. Θα θέλαμε να την επιτύχουμε και συμφωνώ μαζί σας ο καλύτερος τρόπος είναι να υπάρχουν προγράμματα μακροπρόθεσμης διαχείρισης. Τι θα γίνει τώρα. Νομίζω ότι εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε, διότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχουν πολιτικά προγράμματα εν αλλά δεν μπορούμε να τα προχωρήσουμε, γιατί το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν μπορούν να συμφωνήσουν για τις αρμοδιότητές τους. Εδώ είναι παιχνίδι εξουσιών. Ποιος θα αποφασίζει γιατί. Και εντωμεταξύ, όλα αυτά τα πολιετή προγράμματα διαχείρισης έχουν σταματήσει. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα προτείνουμε στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τα πολιτικά προγράμματα διαχείρισης εάν δεν ψηφιστούν. Αυτό έγινε και στο Συμβούλιο φέτος. Στο φετινό Συμβούλιο αποφασίσαμε να προχωρήσουν τα θέματα για κάποια αποθέματα βάσει των μελλοντικών πολιετών προγραμμάτων διαχείριση. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχω και το δικαίωμα να το κάνω κάθε χρόνο αυτό. Σα παρακαλώ λοιπόν βοηθήστε με να ξεπλοκάρει αυτή η κατάσταση γιατί θα είναι φιάλτης και δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση εάν δεν υπάρχουν ε, προγράμματα πολιετού διαχείριση. Για την αλληλεία μικρή κλίμακα. θα του βοηθήσουμε εισαγάγοντα ένα νέο κατόφλι που θα αφορά τη χρηματοδότησή τους. Για την αλία μικρής κλίμακας λοιπόν, από τα ταμεία μας θα δίνεται το 75%. Το 75% της αξίας του προγράμματος. Για την αλληλεία εν γέννη θα έχουμε 50%, αλλά για τη μικρή κλίμακα αλληλεία το ποσοστό θα είναι 75%. Είναι πολύ συγκεκριμένο μέτρο αυτό. Και επίσης θα προσπαθήσουμε να βρούμε και σημεία επαφή με την πολιτική συνοχή. Τώρα με τη νέα νομοθεσία που έχουμε για τη χρηματοδότηση υπάρχουν κάποια νέα προγράμματα από δύο ή τρει γενικές διευθύνσεις τη Επιτροπή και το σκεπτικό μα είναι να έχουμε χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής για τη μικρή κρίμα κασαλία για την ανάπτυξη υποδομών. Όσον αφορά τώρα τα κονδύλια που θα δοθούν στου πλειοκτήτε, δεν θέλουμε να δώσουμε... Ε, χρήματα για νέες ε, μηχανές και νέα μηχανήματα. Υπάρχει τρόπος να εξυγχρονιστούν τα σκάφη. Για παράδειγμα, θα δοθούν χρήματα για αποθηκευτικούς χώρους επί των σκαφών, για νέα ε, εργαλεία αλίευσης ε, ή χρήματα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τους αλληλείς. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε, αλλά δεν θα χρηματοδοτήσουμε κατασκευή νέων ε, μηχανών, γιατί αυτό θα δημιουργήσει υπερβολικές δυνατότητες και τα αλλιεύματές μας θα εξαφανιστούν. Όσον αφορά τα θέματα ελέγχου και τα προβλήματα ελέγχου, ναι, χρειαζόμαστε ένα κανονισμό τον οποίο να μπορούμε να εφαρμόσουμε. Και ήδη υπάρχει βέβαια κάτι, διότι έχουμε το νέο κανονισμό για τους ελέγχους και σε αυτό το νέο κανονισμό για τους ελέγχους λέγεται ότι μπορούμε να έχουμε και μειώσεις για τα αλλιευτικά αποθέματα. Το, αυτό ισχύει και για το σκουμπρί και την ε, υπερβολική αλίευση από πλευράς Ισπανίας. Ε, θα το μειώσουμε, υπάρχει μεγάλη αντίδραση από πλευράς Ισπανίας, αλλά θα εμείνουμε, διότι υπεραλίευσαν πάρα πολύ και πρέπει να κατανοήσουν ότι είναι πάρα πολύ σημαντική συμμόρφωση από πλευράς μας και θα υπάρξει και το ισχυρότερο μας όπλο κατά της μη και αυτό είναι η αιρεσιμότητα. Στη νέα χρηματοδότηση, εάν δεν υπάρχει συμμόρφωση, δεν υπάρχουν και χρήματα. Και αυτό είναι εκ των όνων κάνε φόρος. Και υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο ανέφερε κάποιο συνάδελφο. Εάν ένα κράτο μέλο δεν μα δίνει δεδομένα ή δεν συνεργάζεται όσον αφορά τι επιστημονικέ νομοδοτήσει και πάλι δεν θα δοθούν κονδύλια. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Ιδάλω, ό,τι λέμε δεν θα έχει αποτελέσματα. Για την υδατοκαλλιέργεια. Θα ενισχύσουμε την βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια με ποιο τρόπο. Πρώτον, θα βρούμε νέες περιοχές υδατοκαλλιέργειας μέσω ε, ειδικού ε, χωροταξικού σχεδιασμού για θαλάσσια αποθέματα. Θα υπάρχει και χρηματοδότηση για νέους ανθρώπους που θέλουν να ξεκινήσουν ένα νέο πρόγραμμα υδατοκαλλιέργειας εάν συμμορφωθούν με τους κανόνες ε, βιωσιμότητας. Επίσης θα δώσουμε περισσότερα κονδύλια στα προγράμματα υδατοκαλλιέργειας όταν ε, χρησιμοποιούνται αλλιεύματα ε, τα οποία δεν είναι σαρκοβόρα, ε, όταν δεν χρησιμοποιούνται αλλιεύματα για να χρήσει για ηχθιάλευρα και θα περάσουμε σε εναλλακτικέ λύσεις για τροφή για τα ψάρια ή επίσης θα έχουμε προγράμματα για φύκια και άλλα προγράμματα τα οποία μπορούν να μας δώσουν καλύτερα υλικά για κατανάλωση και όχι μόνο αλλιεύματα. Υπάρχουν νέα προγράμματα και νέα προϊόντα και μπορούμε να τους βοηθήσουμε να ε, έχουν νέα παραγωγή. για το βορρά, το νότο, τις ποσοστώσεις και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται. Ε, κύριε Ρόσμπαχ, νομίζω ότι έχουμε μεγάλες διαφορές εδώ μεταξύ μας. Στη Μεσόγειο δεν υπάρχουν ποσοστώσεις, υπάρχει απλώ ποσόστοση για τον ερυθρό τόνο, δεν υπάρχουν σαφεί επιστημονικέ γνωμοδοτήσει, δεν υπάρχουν κανόνες συμμόρφωση οι οποίοι να είναι τόσο αυστηροί όσο οι βόρειε χώρε και επομένως εδώ υπάρχει ένα κενό το οποίο θα πρέπει με κάποιο τρόπο να πληρώσουμε. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Όσον αφορά τη συμφωνία με το Μαρόκο, ξέρω ότι το ζήτημα αυτό είναι διαφιλονοκόμενο. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειε επ' αυτού διότι θα σπαταλήσουμε πολύ χρόνο. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σεβαστεί την ψηφοφορία του Κοινοβουλίου, υποχρεούμεθα να το κάνουμε και επομένω ε, έχω ήδη καταθέσει μία πρόταση και σήμερα στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος ε, συμφώνησαν επί της προτάσεως αυτής. Θα σταματήσει η αλληλεία εκεί. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας, αφού το Κοινοβούλιο αυτό ψήφισε. Αλλά θα ζητήσω μια νέα εντολή ώστε να καταλήξουμε σε καλύτερη συμφωνία που σημαίνει ότι θα είναι μια συμφωνία πιο φιλική προς το περιβάλλον, ε, μια πιο οικονομικά βιώσιμη ε, και μια συμφωνία που θα βασίζεται στο διεθνές δίκαιο. Είναι ε, πολύ ακαθόδες το ζήτημα αυτό και ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο το οποίο ψήφισε τη συγκεκριμένη σύσταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τόσο μεγάλη πλειοψηφία θα μας υποστηρίξει. Πρέπει βέβαια να πω εδώ ότι θα πρέπει να έχουμε και κατά νου ότι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αυτά τα οποία θα ψηφίσουν στο τέλος. Ό,τι και να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δεν επιθυμούν αυτή τη συμφωνία, τότε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Δαμανάκη διότι μας αναφέρετε τους ακρογωνιαίους λήθους της αλλιευτικής πολιτικής στην Επιτροπή Περιβάλλοντο. Δώσει η Επιτροπή αυτή ε, σας υποστηρίζει διότι είναι σύμφωνα όλα αυτά με τους στόχους μας θα συμβάλλουμε στην νομοθεσία και είμαι πιο πεπισμένος από ποτέ ότι χρειαζόμαστε το άρθρο 50 με την Επιτροπή Αλίας ούτως ώστε να μπορέσουμε ε, να προωθήσουμε τις ιδέες που αναφέρετε εδώ, ούτω ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Καλά Χριστούγεννα, λέει η κυρία Ναμανάκη. Next point, number... Το επόμενο σημείο υπαριθμών 5, οι γυναίκες και κλιματική αλλαγή, γνωμοδότηση ε, της κυρίας Βέβρα Ντεμπρούν. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντεμπρούν με παρακάλεσε να την αντικαταστήσω διότι ε, έχει άδεια λόγω ασθενείας για αρκετό χρόνο και θα ήθελε ο φάκελος αυτός να προχωρήσει, να προωθηθεί παρά την άδειά Να μην χρειάζεται η Επιτροπή να περιμένει την επάνωδό για να έχουμε αυτή τη συζήτηση. Αυτό μου ζήτησε. Οι γυναίκες και η κλιματική αλλαγή είναι κάπως ένα θέμα παρόμοιο με τις αναπτυσσόμενες χώρες και την κλιματική αλλαγή. Οι Γυναίκες, δεν ήσαν ε, τόσο παρούσες μεταξύ ε, αυτών που λαμβάνουν τις αποφάσεις που επηρεάζει την κλιματική αλλαγή. Δεν συμμετείχαν τόσο πολύ στις αποφάσεις, αλλά πολύ συχνά οι γυναίκες υφίστανται τις συνέπειες αυτών των αποφάσεων με σκληρότερο τρόπο. Διαπιστώθηκε εδώ και δέκα χρόνια ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι μόνο θέμα περιβαλλοντικό, είναι θέμα που σχετίζεται με την ανάπτυξη. Και ως θέμα ανάπτυξης έρχεται να προσθεθεί το θέμα των φύλων και οι συνέπειες πάνω στην ισότητα μεταξύ των φύλων. Η τέταρτη έκθεση αξιολόγησης επιβεβαίωσε ότι η επίπτωση της αλλαγής του κλίματος εξαρτάται από την ηλικία, το φύλλο και την κοινωνική τάξη με πιθανότερα θύματα τους φτωχούς. 70% των φτωχών της Ιφιλίου είναι γυναίκες. Σύμφωνα με τις στατιστικές βλέπουμε ότι μεταξύ των ατόμων που χάνουν τη ζωή τους σε θεομηνίες περίπου 85% είναι γυναίκες, περιβαλλοντικοί πρόσφυγες που είναι γυναίκες στο 75%. Και εάν η κλιματική αλλαγή προκαλεί συγκρούσεις, παραδείγματος χάρη γύρω από το είδωρ ή των ε, καλλιεργησίμων εδαφών, οι συγκρούσεις αυτές, οι πόλεμοι των οποίων το δακύβευμα είναι η φυσική πόρη, τότε είναι οι γυναίκες οι οποίες είναι τα πιθανότερα θύματα αυτών των βιαιοτήτων. Σε περιπτώσεις καταστροφών η θνησιμότητα των γυναικών είναι επίσης πολύ μεγαλύτερη. Και Εάν οι ερευνητικές εργασίες λάμβαναν υπόψη το φύλλο, εάν υπήρχε κατανομή των στοιχείων ανάλογα με το φύλλο, θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε καλύτερα τους κινδύνους αυτούς για την υγεία και να θεσπίσουμε προσαρμοσμένα προληπτικά μέτρα. Με άλλα λόγια, είναι επίγουσα ανάγκη να κατανοήσουμε το συντομότερο δυνατόν πώς τα μεταναστευτικά ε, ρεύματα τα οποία προκαλούνται από τις καταστροφές θα μπορούσαν να τύχουν μιας διαχείρισης που να λαμβάνει υπόψη το θέμα του φύλου. Δεν είναι μόνο οι γυναίκες που είναι θύματα, αλλά επίσης ε, αυτό που είναι σημαντικό είναι οι γνώσεις που έχουν οι γυναίκες. Πολύ συχνά η ενημέρωση, οι παραδοσιακές γνώσεις ο τρόπος ο παραδοσιακός δράσης που προκαλεί ε, ε, λιγότερες εκπομπές ε, και ζημιές είναι οι γνώσεις που έχουν οι γυναίκες και που τις μεταβιβάζουν. Τις μεταδίδουν κάτι που συχνά το ξεχνούμε η προοπτική ανδρών γυναικών μέσα στη συζήτηση για το κλίμα είναι κάτι το πάρα πολύ ε, εύστοχο και προσωπικά ε, θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτά που προτείνει ε, η συγγήτρια στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Θα ήθελα εγώ προσωπικά να προσθέσω ότι το σημαντικότερο από την άποψη των γυναικών και από την άποψη όλων θα πρέπει να αλλάξουμε την κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι το σημαντικότερο για όλους. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη σε όλα τα επίπεδα τις γυναίκες και όταν θεσπίζουμε μέτρα προσαρμογής θα πρέπει να μεριμνήσουμε όλα αυτά να μην θίξουν περισσότερο την κατάσταση των γυναικών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπουμε πώς και στον Ντάρμπαν και αλλού το θέμα αυτό ε, συνδέεται, πώς συνδέεται ο ρόλος των γυναικών με την κλιματική αλλαγή. Στην γνωμοδότησή μας ε, στην Επιτροπή Γυναικών στο Κοινοβούλιο, το λάβαμε αυτό υπόψη, υπάρχουν, ε, θέλει κανείς να λάβει τον λόγο, παρεμβάσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Ντεμπρούν διότι νομίζω αυτή η γνωμοδότηση είναι πάρα πολύ εύστοχη. Θα ήθελα και εγώ να ζητήσω να προσθεθεί κάτι σχετικά με τον σημαντικό, τον κρίσιμο ρόλο των γυναικών στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Και συνεπώς θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη ευρύτερης και μια ε, διπλωματίας, κλιματικής περιβαλλοντικής διπλωματίας σε όλες τις διαπραγματεύσεις. Μιλήσατε κύριε Πρόεδρε για το Durban. Μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα με την εισαγωγή της αντίληψης της ήπιας δύναμης στην κλιματική διπλωματία στις ε, διεθνείς διαπραγματεύσεις περί κλίματος, διότι πριν από δέκα μέρες, όπως άκουσα, ε, ο πρόεδρος ε, της διάσκεψης ζήτησε από την κυρία Κόνι Χίλντεγκαρντ, την επίτροπό μας και στον Υπουργό Εξωτερικών της τον Υπουργό Περιβάλλοντας, με συγχωρείτε, της Νοτιού Αφρικής να βρουν μια λύση σχετικά με την Ινδία σε 10 λεπτά και διαπραγματεύτηκαν μαζί οι δύο γυναίκες και μπόρεσαν να επιτύχουν ένα συμβιβασμό όχι σε 10 λεπτά αλλά σε 15 λεπτά. Μπορούμε λοιπόν την αντίληψη αυτή της ήπιας δύναμης να την χρησιμοποιήσουμε, διότι χρησιμοποιείται και σε άλλες, στη διπλωματία γενικά και όχι μόνο στην διπλωματία την κλιματική. Τονίζω την σημασία των γυναικών για την εφαρμογή μέτρων μετρίασης στην καθημερινή ζωή, εξοικονομώντας ενέργεια με μέτρα ανακύκλωσης και με την χρήση φιλικών και βιολογικών προϊόντων και θέλω να τονιστεί η σημαντική συμβολή των γυναικών που μπορούν να επιφέρουν καινοτομίες ε, τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στα νοικοκυριά. Θα πρέπει να καλέσουμε τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών να ε, εισαγάγουν την αρχή της κλιματικής δικαιοσύνης διότι πρέπει να επιμείνουμε ότι υπάρχει μεγάλη αδικία στο θέμα της κλιματικής αλλαγής που έχει δυσμενείς επιπτώσεις πάνω στις φτωχές χώρες και στις γυναίκες ειδικότερα. Και θα πρέπει να αξιολογήσουμε μέχρι ποιου βαθμού οι πολιτικές που σχετίζονται με το κλίμα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των γυναικών και, τις καλούν, και τους καλούν να λάβουν υπόψη την ισότητα των φύλων στις πολιτικές αηφόρου ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Πλάμ για αυτές τις παρατηρήσεις. Δεν νομίζω ότι κανείς άλλος θέλει να λάβει τον λόγο. Η προθεσμία ε, για την κατέθεση των τροπολογιών είναι αύριο στις 12. Αυτό είναι απαραίτητο για την λήψη αποφάσεως στην Επιτροπή Γυναικών. Φτάνουμε τώρα στο σημείο 6 σχετικά με την απαλλαγή. Πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η συγκητής είναι ο Κρεσένσο Ριβελίνη και σήμερα αντικαθίσταται από την Ελίζαμπέτα Γκαρντίνη. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρου του κυρίου Ριβελίνη, αλλά σήμερα δεν ε, μπορούσε να παραστεί τη συγκεκριμένη ώρα. Γι' αυτό λοιπόν μου ανέθεσε να ακούσω τουλάχιστον τις υποδείξεις των συναδέλφων. Έχουμε εδώ ένα περίγραμμα της γνωμοδότησης. Δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι θα πρέπει να το διατρέξουμε λίγο από κοινού. Είναι έξι μόνο και τα σημεία όπου αναφέρονται κάποια στοιχεία τα οποία θεωρούνται θετικά και προτείνεται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να υπάρχουν κάποια κριτήρια κατά νου ε, και να ληφθούν δεόντω υπόψη. Στο σημείο 1 υπογραμμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να δεσμευτεί στη χρηματοδότηση προγραμμάτων που θα πληρούν αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια προωθώντα μια βιώσιμη ανάπτυξη. Στο σημείο 2 εκφράζεται ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανέβασε στα 19 δισεκατομμύρια ευρώ, επομένως ε, ε, κατά 30% τη πιστώση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις επενδύσεις που προβλέπονται για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων υπέρ του κλίματος, τα οποία αφορούν τομείς όπως ε, η ενεργειακή απόδοση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι μεταφορές και Στο τρίτο σημείο καλείται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να δεσμευτεί να μην χρηματοδοτεί σε αυτή την περίπτωση κάποιου τύπου προγραμμάτων, προσδιορίζοντα απαγορευμένε ε, ζώνε και απαγορευμένε τεχνολογίε. Στο τέταρτο σημείο εκφράζεται ικανοποίηση για την υποστήριξη εκ μέρου τη ΕΤΕΗ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και ε, λέγεται ότι περάσαμε από κατά 6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2010 στα ε, συγγνώμη, από 500 εκατομμύρια ευρώ το 2006 στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2010, στο πέμπτο στοιχείο εκφράζεται ικανοποίηση για το γεγονός ότι ε, βελτιώθηκε η τεχνική και εσωτερική συνιστότητα και χρησιμοποιούνται πυροχνόμοντες που εργάζονται κατά πρώτο λόγο σε προγράμματα ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών. Και τέλος, το 6, ζητάτε από την Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα Επενδύσεων να θέτει αυστηρούς όρους για τα προγράμματα παραγωγής ενέργειας τα οποία βασίζονται στον άνθρακα και στο λιγνίτη διότι θεωρείται ότι με την εφαρμογή αυτών των κριτηρίων θα έχουμε μια ταχεία κατάργηση της στήριξης της τράπεζες, στην παραγωγή παραγωγή ε, για υψηλές εκπομπές άνθρωπα. Αυτά είναι τα σημεία της γνωμοδότησης. Και εγώ θα μεταφέρω στο συνάδελφο όλα τα σχόλια των ε, παρισταμένων. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και η ομάδα μου χαιρετίζει το σχέδιο αυτό της γνωμοδότησης του κ. Ριβελίνη. Μας φαίνεται ότι είναι αρκετά ισορροπημένο. Αναφέρονται μια σημαντικά σημεία. Μας αρέσει η γνωμοδότηση όπως είπα σημειώνουμε τους ε, δείκτες ε, χρηματοδότησης της ΕΤΕΠ όσον αφορά τα σχέδια που σχετίζονται με το κλίμα, από αποτελεσματικέ ενέργεια, ανενώσιμες πηγές ενέργειας και προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές. Επίσης, μας άρεσε η ιδέα που εξετάζονται οι λεγόμενες απαγορευμένες ε, τεχνολογίε. Έχουμε έναν μαύρο κατάλογο, όπω λέμε. Ίσως κανένα θα μπορούσε να εισαγάγει και μία σειρά παραδειγμάτων τέτοιων σχεδίων που απογραφτήκαν ή που δεν ενεκρίθησαν. Δεν πρέπει να φοβούμαστε τον να κατανομάζουμε και να ντροπιάζουμε σε αυτόν τον τομέα, γιατί πολλές φορές αυτού του είδους τα σχέδια επαναλαμβάνονται μετά σε άλλες χώρες. Θα θέλαμε μάλιστα να προχωρήσουμε περισσότερο και να έχουμε και μια σειρα παρεδειγμάτων τετοιων σχετίων που απογραφτηκαν η που δεν ενεκριθησαν δεν πρεπει να φοβουμαστε το να κατανομαζουμε και να ντροπιαζουμε σε αυτον τον τομεα γιατι πολλέ φορες αυτου του είδου τα σχεδια επαναλαμβανονται μετα σε άλλε χώρε. θα θελαμε μαλιστα να προχωρησουμε περισσοτερο και να εχουμε και μια θεα ενα φε, κατάλογο. Όπως παραδείγματο χάρη είναι αυτές οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στο μεθόριο αν θέλετε όπως ε, καύση απορριμμάτων κλπ. Η... Ξέρουμε ότι γίνονται οι έρευνες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων για τα σχέδια αυτά. Αλλά ίσως μπορούσε κανένας να κάνει κάτι παραπάνω, να κάνει ε, στρατηγικές περιβαλλοντολογικές αξιολογήσεις. Θα πρέπει η ΕΤΕ να εξετάσει που ενδεχομένως μειώθηκαν τα εθνικά πρότυπα για να γίνουν δεκτά κάποιες, κάποια τέτοια προγράμματα που βρίσκονται στο μετέχνιο. Ξέρετε την εικόνα αυτή την ε, μαμούδων που κλείνουν τα μάτια στα αυτιά τους και το στόμα τους και δεν λένε τίποτα, δεν ακούν τίποτα, δεν βλέπουν τίποτα και αφήνουν να γίνουν τα πάντα. Τέλος, θα ήταν ε, ίσως ενδιαφέρον ένας άλλος τομέας για τις ε, ε, νότιες χώρες μέλη που βρίσκονται στα παράκτια της Μεσογείου το θέμα της διαχείρισης των υδάτων. Εκεί θα πρέπει να γίνει κάτι παραπάνω νομίζω. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ζαμχοντή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον ε, κύριο Ριβελίνη και την κυρία Γαρδίνη που προετοίμασαν αυτό το προσχέδιο και μας το παρουσιάζουν εδώ. Μόλις ήρθα μάλιστα από την Επιτροπή ε, Ελέγχου του Προπολογισμού που ο πρόεδρος μάλιστα παρουσίασε την ετήσια έκθεση και είχα την ευκαιρία να του υποβάλω κάποιες ερωτήσεις γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένο με τις εξελίσεις μέσα στα πλαίσια Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το περιβάλλον. Διπλασίασαν σχεδόν τα σχέδια από 10 σε 19 δις ευρώ σε 2-3 χρόνια. Είναι πάρα πολύ θετική αυτή η εξέλιξη. Ομολογώ όμως επίσης ότι φαίνεται ότι η συγκέντρωση γίνεται κυρίως στα θέματα κλίματος και θα ήθελα να να σας πω ότι ρώτησα τον κύριο Μάιστατ, αναγκάστηκα όμως να μην ακούσω την απάντησή του, γιατί βιαζόμουν να έρθω εδώ και εκείνος έτσι και δεν μπορούσε να απαντήσει όλες τις ερωτήσεις. Ρωτώ λοιπόν, μήπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν θα θέλει να συγκεντρώσει λίγο στην προσοχή σας περισσότερο στην αποτελεσματική χρήση των πόρων, φυσικών πόρων και επίσης όσον αφορά την βιοποικιλομορφία. Μια από αυτά είναι από τα πιο μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και λείπει από την ετήσια έκθεση. Τέλος τον επέκρινα, γιατί παρόλο που είναι ένα τμήμα μόνο των σχεδίων του ΕΣΕΤΕ, θα πρέπει να επενδύνουμε λιγότερο στα, ε, στις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα. Παρόλο που είναι μόνο το 10% θα πρέπει να ε, πιστήσουμε την προσοχή στην ΕΤΕΠ να μην χρηματοδοτεί αυτά τα σχέδια στο μέλλον. Ευχαριστώ. Τώρα το σας ευχαριστώ. Κάποιος άλλος δεν θέλει το λόγο. Όχι. Ωραία. Ο κύριο Καράνο, παρακαλώ. Της, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστώ τον εισηγητή του κύριο Ριβελίνη για την ομοδότησή του. Και να ευχαριστώ και, ευχαριστήσω και για τις ερωτήσεις που μας υπευρύθησαν. Ε, Σημειώσαμε όλες τις ε, προτάσεις και συστάσεις που υπάρχουν στην χρωμοδότηση αυτή. Ιδίως ε, είδατε ότι η τράπεζα πιέζεται ώστε να γίνει μια πλήρη περιβαλλοντική τράπεζα όπως αποδεικνύονται και από τα στοιχεία που υπάρχουν όσον αφορά για τους καταλάβους, αυτούς μαύρους, τους θεούς, είναι κάτι που ήδη γίνεται στην ΕΤΕ να χρησιμοποιεί δηλαδή πλήρως τα πρότυπα των ε, οδηγιών και πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο εσωτερικό της Ένωσης, αλλά και κατά δυνατόν να εφαρμόζονται τα ίδια κριτήρια και εκτός της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προστατεύεται η ποικιλομορφία παντού. Να τηρείται το Natura 2000 κλπ. Το ίδιο ισχύει και για τα φράγματα. That we finance, uh, although... ε, παρόλο που θα πρέπει να σημειώσετε ότι μέσα στα πλαίσια των συμφωνίων εταιρικής σχέσης και ε, τη συμφωνία Κοτονού λαμβάνουμε υπόψη μας όλες τις πηγές που αφορούν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. και όλα αυτά που σχετίζονται με τα φορολογικά εισοδήματα και τις δεσμεύσεις που υπάρχουν, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρους παρουσίαση προς την Κομισιόν για του τα χρήματα που χρησιμοποιούνται και που μένουν στη χώρα αυτή λόγω των επενδύσεων. Ε, επίσης, έχω να πω ότι για την ενέργεια χρηματοδοτούμε το κατά 75% ανανόσιμες πηγές ενέργειας. Και έχει μειωθεί η χρηματοδότηση ορυκτών ε, πηγών ενέργειας κατά 10%. Και μόνο εκεί που κάτι τέτοιο δικαιολογείται από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της ε, κάποιου κράτου που έχουν μια πολιτική να βασίζονται σε αυτού του είδου τις ε, προοδεσίλες, όπως στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη. Παραδείγματο χάρη, όταν χρηματοδούμε ε, μονάδες παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, ε, χρησιμοποιούν πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια περιβαλλοντικής προστασία, Παραδείγματο χάρη να χρησιμοποιείται η βέλτιστη δυνατή τεχνολογία ή να ε, είναι οι μονάδες αυτές ε, στο μετέχνιο πραγματικά της καινούργια τεχνολογίας και να ελέγχονται όλες οι εκπομπές. Να μειώνεται το δεξιό του άθρακα και όχι να αυξάνεται. Τέλος, αναφορά τα πρότυπα που χρησιμοποιούμε, έχω να τονίσω ότι αυτό ε, στον τομέα ακριβώς αυτό για τα δικτά καύσιμα έχουμε διαγράψει 20% σχέδια. 20 περιπτώσεις δηλαδή σχεδίων που υποβλήθησαν στην τράπεζα δεν έλαβαν χρηματοδότηση γιατί δεν ήταν σύμφωνα με τις πολιτικές μας. Και είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πρόταση για βελτίωση του πολιτικών μας αναθεωρήσαμε συγγνώμη, τα πρότυπα μας το 2009 μετά από διαβούλευση και από το Κοινοβούλιο και ευχαρίστω θα σας ακούσουμε τις προτάσεις σας για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Είμαστε η Τράπεζα Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι στο να εφαρμόσουμε τις πολιτικές ε, που έχουν περάσει από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μήπως ο εισηγητής θέλει να λάβει και πάλι το λόγο. Όχι. Όχι. Σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι 20 ε, Δεκεμβρίου στις 18 ε, η ώρα. Θα περάσει αυτό από την Επιτροπή στις ε, ελέγχου του προϋπολογισμού στις 29 Φεβρουαρίου. Τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το 7, επαλλαγή γενική για τον προϋπολογισμό. Κυρία Γιούτα Χόγκ είναι η συγγήτριά μας. Κυρία Χόγκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. έχουν φτάσει στην ήπια ε, δύναμη αλλά με σκληρά στοιχεία. Λοιπόν, οι προτάσεις μου για την απαλλαγή υπέβλησαν σχετικά έγκαιρα ούτως ώστε να τηρούνται όλοι οι όροι για την σωστή μετάφραση των κειμένων αυτών. Ξέρω ότι υπάρχουν ήδη επικρίσεις όσον αφορά την προθεσμένη υποβολή τροπολογιών η οποία λύγει αύριο στις 6 το απόγευμα. Αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα. Γιατί ακριβώς πρέπει έγκαιρα να ε, εγκρίνουμε δική μας πρόταση, ούτως ώστε η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού που είναι επί της ουσίας αρμόδια για την απαλλαγή, να έχει στα χέρια της την γνωμοδότησή μας όταν ψηφίζει. Και η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού με επιστολή του Προέδρου και της ηγήτριας για τις υπηρεσίες είπε για άλλη μια φορά ξεκάθαρα ότι χρειάζεται τη δική μας γνωμοδότηση πριν από τις 22 Φεβρουαρίου. Και αν κοιτάξετε το χρονοδιάγραμμα, αφαιρέστε τις διακοπές για τα Χριστούγεννα, βλέπετε ότι δεν έχουμε άλλη λύση παρά αύριο το απόγευμα στις 6 να λύγει η προθεσμία για τις τροπολογίες που θα πρέπει να τις έχουμε υποβάλει μέχρι τότε όλες. Δεν θέλω να σας γκρινιάζω, αλλά κοιτάω γύρω μου. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι πολλοί συνάδελφοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν τροπολογίες. Γιατί όσο έντονη είναι η συμμετοχή κατά δυνατόν για τη συζήτηση, ε, τόσες θα έχουν θα είναι και οι υποβληθείς της Τώρα, άμα κοιτάξουμε το προπολογισμό μας και γενικά τον προπολογισμό για την Επιτροπή Περιβάλλοντος, όλο το τομέα, δηλαδή περιβάλλον, δημόσια υγεία και ασφάλεια τροφίμων, αν το κοιτάξουμε αυτό, βλέπουμε ότι είμαστε αρμόδιοι για 0,76% του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Δηλαδή δεν είμαστε υπεύθυνοι ούτε για το 1% του προπολογισμού. Ξέρω βέβαια ότι μια σωστή περιβαλλοντολογική πολιτική μόνο παρεμπιπτόντως έχει σχέση με οικονομικά. Γιατί αυτή η πολιτική περιβάλλοντας δημόσιας υγείας και ασφάλειας τροφίμων σχετίζεται κυρίως με νομοθεσία. Ε, το κάνουμε αυτό. Και λέω στους αδέρφους, και θα ήθελα αυτοί που είναι παρόντες να το πούνε και στους άλλους, να ενθαρρύνουμε όλους να εμπλακούν σε εκείνους τους τομείς όπου μπορεί επίσης να εφαρμοστεί η περιβαλλοντική πολιτική. Ένα παράδειγμα είχαμε προηγουμένω παρουσία της Επιτρόπου Δαμαδάκη όταν ζητήσαμε για την ε, πολιτική αλίας. Εάν εμείς ως Επιτροπή Περιβάλλοντος δεν εμπλακούμε εκεί, το ίδιο ισχύει για τη μεταρρύθμιση της αγροτικής πολιτικής. Εάν δεν το κάνουμε, εγκαταλείπουμε έναν τομέα σημαντικό στον οποίο θα μπορούσαμε να παρέμβουμε περιβαλλοντολογικά. Σας παρακαλώ, αναμειχθείτε στα πάντα. Και ξέρετε ότι εάν δεν κάνουμε τίποτα μέχρι του χρόνου θα παραμείνει μέχρι το 2020. Με όλο το δημοσιονομικό πλαίσιο. Τότε ο Επιτροπή σου, ξέρω αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ε, απαλλαγή, αλλά θέλω πραγματικά να ταρακουνήσω, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, του συναδέλφου. Στην Επιτροπή σου, λοιπόν, παλιά είχαμε ορίσει τάσει και ε, άγουσε πώ θα μπορούσαμε, κατά τη γνώμη μα, να δούμε μια μεταρρύθμιση των πολιτικών τους ώστε να είναι πιο βιώσιμες, περιβατολογικές, ε, να μειώνουν το δεξίο του άνθρακα. Και έτσι να βοηθήσουμε γενικά να καταπολεμηθεί η αλλαγή κλίματος. Και παρακαλώ, παρακαλώ, ασχοληθείτε με αυτό ξανά και ξανά και ξανά. Τελεία. Τα άλλα μπορείτε να διαβάσετε άμα θέλετε. Σε γενικές γραμμές δηλαδή μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με το ποσοστό εκτέλεσης για το 2010 της Γενικής Διεύθυνσης για το κλίμα, για το περιβάλλον και για την ΣΑΝΚΟ. Μπορούμε σε γενικές γραμμές λέω να είμαστε ικανοποιημένοι με τα στοιχεία που μας δίνουν. Προσπάθησαν πολλά να κάνουν σωστά, καλά, και το μόνο πραγματικά παρεμβατολογικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα LIFE, ε, πραγματοποιήθηκε πολύ καλά. Διαφορετικά από το όπως ε, προβλέπετε αρχικά, ξέρετε ότι υπήρχαν ενδεικτικές ε, αναφορές για τα κράτη-μέλη και μόνο αν υπήρχε έλλειψη αιτήσεων από τα κράτη-μέλη ή της ποιότητας των αιτήσεων θα μπορούσαν τα χρήματα αυτά να δουν σε άλλες χώρες μέλη η Κομισιόν ή και κάποιες διοικήσεις κρατών μελών θα πρέπει να εξετάσουν πού μπορούν να υπάρχουν βελτιώσεις. Τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας, μάλλον που διαθέσαμε, χρησιμοποιήθηκαν κατά πολύ διαφορετικούς τρόπους. Αν το συζητήσουμε αυτό, ότι τα χρήματα που διαθέθηκαν, αυτά που προβλέπονται δηλαδή στο προπολογισμό, και εκείνα που δαπανήθηκαν μετά δεν συμφωνούν μεταξύ τους τα δύο ποσά αυτά. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διάφορα αιτία. Ζωκτονίες παραδείγματος χάρη ε, δεν υπήρχαν τόσες ασθένειες, δεν χρειαζόμασταν συμπληρωματικά μέτρα, δεν χρειαζόμασταν ε, προγράμματα εμβολιασμού και δεν χρειαζόταν να αγοράσουμε ε, υλικό για το εμβολιασμού. Αλλά βέβαια τα ποσά ήταν κάπως υψηλά για τις επιζωτίες αυτές. Θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο ανοιχτοί, πολύ πιο σαφείς. Γιατί ξέρουμε όταν η ΣΑΜΚΟ λέει κάτι στη Γενική Διεύθυνση για τον προπολογισμό ή τι θα πρέπει να προβληθεί, προβλεφθεί, Εάν θα τώρα απομένουν τόσα χρήματα, παρά στις σπάθιες ακρίβειας που έχουν γίνει, θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο ακριβείς. Πάντως εγώ δεν μπορώ παρά να συστήσω να δώσουμε την απαλλαγή αυτή στις Γενικές Διευθύνσεις ε, ΣΑΝΚΟ, Περιβάλλον και Κλίμα. Άμα δούμε τώρα τις ε, υπηρεσίε για τι οποίε είμαστε υπεύθυνε. Περιβάλλοντο στην Κοπενχάγη, χημεία στο Ελσίνκι, ε, φαρμακευτικά προϊόντα στο Λονδίνο, κέντρο για την πρόληψη ασθενειών στην Στοκχόλμη και υπηρεσία για την ασφάλεια τροφίμων στην Πάρμα. Αυτές είναι οι υπηρεσίες τις οποίες εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Για τις τέσσερις πρώτες, δεν χρειάζεται νομίζω να τις ξανασυζητήσουμε. μπορούν να συστήσουν την απαλλαγή χωρίς περιορισμούς. Και βλέπουμε ότι η υπηρεσία περιβάλλοντος εργάστηκε πολύ καλά, δαπάνησε τα χρήματα ακριβώς όπως τα προβλέψαμε. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι η υπηρεσία περιβάλλοντος θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω όσον αφορά την επικοινωνία. αλλά ήδη έκανε κάποιες προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή για το 2011 χωρίς να πούμε ότι χρειάζεται να κάνει κάτι παραπάνω και νομίζω ότι η κατάσταση βελτιώνεται συνεχώς. Λοιπόν, όσον αφορά την επικοινωνία και την δημόσια αντίληψη το τι κάνει η υπηρεσία αυτή, δεν πρέπει να ανησυχούμε περαιτέρω. Το ίδιο μπορούμε να πούμε για την υπηρεσία για την χημεία, που όχι το 2010, όπου αναγκαστήκαμε να μεταβάσουμε κάτι πάνω από 33 εκατομμύρια από τον κοινοτικό προπολισμό. Φέτος όχι. Χρηματοδοτήθηκε απόλυτα από τις εισφορές. Αλλά θα πρέπει να πούμε επίσης ότι μετά που ξεκίνησε η κανονική εργασία στην υπηρεσία αυτή χημίας, ε, έκανε μια σειρά δράσεων όσον αφορά την ε, επικοινωνία, όσον αφορά στο σελίδε, ε, ε, μέρες, ε, ημερίδες ενδιαφέροντος και ούτω καθεξής, ούτως ώστε ενημερώθηκε καλύτερα η κοινή γνώμη το τι κάνει αυτή η υπηρεσία και ταυτόχρονα όλοι εκείνοι που έπρεπε να καταγράψουν τις, τα προϊόντα τους εκεί είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν καλύτερα έχοντας παρακολουθήσει τα σχετικά και κλπ. Λοιπόν, δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτή. Η αίμα που ε, στο Λονδίνο η οποία ήταν κάπως ε, ανησυχητική στην αρχή το ηλεκτρικό συνέδριο δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένο ακόμα με τα θέματα της ε, πληροφορικής εκεί αλλά δεν μπορεί κανένας να κάνει κάτι ξαφνικά Ε, και βλέπουμε ότι λεπτομέρειες στον αφορά και οι συμβάσεις για την πληροφορική έχει βελτιωθεί. Αυτό που θα πρέπει ακόμα να, περισσότερο να βελτιωθεί και ελπίζω ότι αυτό θα το δούμε από την επόμενη μελέτη που έχουμε αναθέσει ως Επιτροπή Προπολογισμού είναι ότι εμείς χρειάζεται πάντα να ε, χρηματοδοτήσουμε την ΕΜΑ. Ε, αυτή η υπηρεσία όμως για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι εθνικές υπηρεσίες είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν και μάλιστα σημαντικά ποσά. Δηλαδή εθνικές υπηρεσίες χρηματοδοτούν κατά 50% και παραπάνω από την αίμα, δηλαδή από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν ε, αυτό που είχαμε φανταστεί αρχικά. Πάντως ε, μέσα στα πλαίσια της ε, δημοσιονομικής ε, διαδικασίας και της διαδικασίας απαλλαγής αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σχετικό. Θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε και να δούμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται και τι γίνεται με τις πληρωμές προς τις εθνικές αυτές υπηρεσίες. Τέταρτη, στο Χόλμη. έχω, όχι να γκρινιάξω, αλλά πώς να σας το πω. Μια που μία από τις αρχές ε, του προπολογισμού μας είναι ότι στους χαρακτήρας, είναι δύσκολο να πρέπει να, να εκτιμήσει κανένας πόσα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν σε ένα χρόνο. και το 2010 υπήρχε σημαντικό πλεόνασμα στην υπηρεσία αυτή. Συνήθω κανένα χαίρεται να έχει πλεονό, πλεόνασμα άμα δεν ε, χρειάζεται να βάλει χρέη. Αλλά λόγω του τίσου χαρακτήρα του προπολισμού είναι αυτό προβληματικό. Η κατάσταση βέβαια βελτιώθηκε κάπως και το 2010 Το θέμα είναι ότι η υπηρεσία αυτή ανέβαλε την μετακόμιση σε ένα νέο κτίριο. Κατά τα άλλα και όσον αφορά αυτή την υπηρεσία στο Στοκόλμη, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι πρέπει να βελτιώσει κάποιες διαδικασίες. Ναι, τώρα θα μπορούσε κανένα να πει εντάξει. Ω συνήθω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο βορρά πάνε καλά τα πράγματα, στο νότο τσίρκο. Ναι, στην Πάρμα φτάνω. Και υπάρχουν πάλι προβλήματα. Η ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων του Οργανισμού Αυτού Ασφάλειας μα, στην Πάρμα που έχει διαφυσβητηθεί, επικριθεί, δεν ξέρω πώ θα το πείτε αυτό. Παίζει ρόλο και στη διαδικασία απαλλαγή 2010. Πρέπει βέβαια να διακρίνει κανένας ανάμεσα στην ανεξαρτησία των επιστημονικών επιτροπών και που, πώς καταλήγουν στο περιεχόμενο των ε, εκτιμήσεων τους οι επιτροπές αυτές και από την άλλη μεριά τους συνεργάτες που φεύγουν από την ΕΦΣΑ, από την Επιτροπή Ασφάλειας ε, Τροφίμων και πάνε σε μια επιχείρηση μετά. Ε, σε επιχειρήσεις οι οποίες αφορούνται από αξιολογήσεις και εκτιμήσεις της ΕΦΣΑ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει βέβαια κανονισμός για το προσωπικό, όπου κατά βάση διακανονίζεται αυτό. Αυτό που θα πρέπει να κάνουν αυτές οι υπηρεσίες είναι να εφαρμόσουν αυτό το άρθρο του κανονισμού προσωπικού στη δική τους περίπτωση. Όσο γίνεται. Και ακριβώς είχαμε μία υπόθεση όπου μία ε, συνεργάτης ε, της, ε, ΕΦΣΑ πήγε στην εταιρεία Συγγέντα είναι μια επιχείρηση που παράγει με τη βοήθεια γενικά τροποποιημένων οργανισμών. Και αυτή η λεγόμενη φάση ε, cooling off, δηλαδή ανάμεσα στην εγκατάλειψη της θέσης στην ΕΦΣΑ και στην, εισαγωγή, στην είσοδο μάλλον στην επιχείρηση, αυτή η περίοδος δεν τηρήθηκε. Και αυτή η συνεργάτης έχει και στη Σιγέντα ακριβώς τον ίδιο τομέα με τον οποίο ασχολείται όπως και στην ΕΦΣΑ. Πρέπει βέβαια να μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι 19 Δεκεμβρίου, το θέμα ξεκίνησε στις 8 Δεκεμβρίου και υπάρχει αλληλογραφία εν τω μεταξύ εγώ δεν μπορώ να πω σήμερα οριστικά τίποτα αλλά θέλω να πω ότι σε αυτό που μεταβιβάζουμε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού Δεν συμπεριλαμβάνεται μια δική μου τροπολογία, στην οποία αναφέρω ότι τώρα αμέσως αποφασίστηκε νομίζω 15 Δεκεμβρίου. Θα πρέπει, λέω, η ΕΦΣΑ επιτέλους να εφαρμόσει τους κανόνες του κανονισμού προσωπικού. Ε, βέβαια, δεν άρχισαν στις 8 Δεκεμβρίου να το σκέφτονται και στις 15 το εγκρίναν αυτό. Η διαδικασία ήταν αρκετά πιο γορονοβόρα. Πέρασαν δύο χρόνια όμως. Είναι κάπως πολύ χρόνος αυτός και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να προτείνουμε να... αυτή την τροπολογία και ταυτόχρονα προσπαθήσουμε να καλέσουμε την Κατρίν Λέν και να την ερωτήσουμε για την υπόθεση αυτή. Τίποτα άλλο δεν θυμάμαι να έχω να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Θα αλλάξω καπέλο τώρα για να λάβω τον λόγο εκ μέρους ε, του σκιώδους εισηγητού της ομάδας Άλντε ε, και θα, κύριο Παναγιώτη και επίσης ε, θα μιλήσω και προσωπικά. Ο κύριος Παναγιώτοφ θα ήθελε να σας συγχαρεί για την εργασία σας για τον προϋπολογισμό. Θα ήθελα να επισημάνει ορισμένα σημεία. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ρωτήσει όταν ε, με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού θα έχει τεθεί η ατζέντα. Θα, ε, ε, θα πρέπει η Επιτροπή ΕΜΒΗ να έχει αρκετό χρόνο για να αναλύσει τα στοιχεία όχι μόνο για την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου που προβλέπεται για την αρχή του Φεβρουαρίου 2012, αλλά και για άλλες εκθέσεις ε, της ε, Γενικής Διεύθυνσης ε, της Επιτροπής. Δεύτερον, λαμβάνοντας υπόψη τους ελέγχους του ελεγκτικού ε, συνεδρίου για τις συγκρούσεις συμφερόντων στην ΕΦΣΑ ε, και στην Επιτροπή Φαρμάκων. Ο κύριος Παναγετόφ θα ήθελε να αναβάλει την απαλλαγή μέχρι ότου οριστικοποιηθεί έκθεση. Ο κύριος Παναγιωτόφ θα προτείνει τροπολογίες ζητώντας από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό ε, Συνέδριο περισσότερο έλεγχο απόδοσης για να έχουμε μια καλύτερη γενική εικόνα σχετικά με την διαχείριση των οργανισμών. Εγώ προσωπικά θα καταθέσω τροπολογία για την αναβολή της απαλλαγής τόσο για τον Οργανισμό Φαρμάκων όσο και για την ΕΦΣΑ. Όσον αφορά την αίμα, όπως ξέρετε, αυτός ο οργανισμός ήδη ήταν στο στόχαστρο του Κοινοβουλίου στην αρχή του έτους, εφόσον είχαμε αναβάλει την απαλλαγή κατόπιν προτάσεως της Κόκομπου. Μεταξύ των αιτιάσεων ήταν η διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων των εμπειρογνωμόνων που είχαν εμπλακεί στην αξιολόγηση των φαρμάκων και την περίπτωση των revolving doors του πρώην διευθυντή. Όσον αφορά τώρα τη σύγκρουση συμφερόντων, στο ψήφισμα σχετικά με την τελική απόφαση για το 2009, το Κοινοβούλιο είχε δώσει την απαλλαγή για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, λόγω των απαντήσεων του οργανισμού σχετικά με την τήρηση του διοντολογικού κώδικα και δεύτερον, περιμένοντας να εφαρμόσει Τη της συστάσεις. Ο οργανισμός άρχισε μια πολιτική διαφάνειας για τις συγκρούσεις συμφερόντων των εμπειρογνωμόνων που ήταν στις ομάδες. Πολύ καλά. Αλλά αν δεν επαληθεύσουμε όλα αυτά, αυτό είναι ευσεβής πόθος. Είχαμε, ε, πόθος. Ήταν, είχαμε μια παλιά συζήτηση εδώ, Μισελ Ριβαζή θυμάται, για την επαλήθευση των δηλώσεων. Στην τελική ψηφοφορία της τελευταίας απαλλαγής είχαμε δεχθεί το επιχείρημα του οργανισμού που έλεγε ότι δεν αναπόκειται σε αυτό να επαληθεύσει τις δηλώσεις των εμπειρογνωμόνων διότι αυτό είναι έργο των αρμοδίων αρχών των κρατών μέλων. Πολύ καλά, αλλά ίσως η θα μπορεί να δει ποιοι είναι οι συγκρούσεις συμφερόντων και οι αιτιάσεις που έχουν κατατεθεί. Ε, και αυτό είναι ανησυχητικό. Εγώ προσωπικά αν η αίμα, εφήρμοσε τις συστάσεις και διαπίστωσα δύο πράγματα. Πρένοντας ένα δειγματολόγιο Γάλλων εμπειρογνωμόνων που δουλεύουν στην ΕΠΣ, συνέκρινα τις ετήσιες δηλώσεις που είχαν κατεθέσει στην ΕΜΑ και στον Γαλλικό Οργανισμό. Και είδα αρκετές διαφορές. Πολλές φορές παραλήψεις στις δηλώσεις στην ΕΜΑ. Δεύτερον, σε πάρα πολλές περιπτώσεις ε, δεν υπάρχει καμία δήλωση στην ΕΜΑ εκ μέρους των εμπειρογνωμόνων, ενώ στην Γαλλία αυτά δηλώνονται. Τρίτον, πήρα ένα δείγμα μερικών μελών ε, της Διαχειριστικής Επιτροπής και ένας παρέλειψε να αναφέρει τις σχέσεις με την φαρμακευτική βιομηχανία, ενώ οι κανόνες της ΕΜΑ λένε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι σχέσεις μέχρι πέντε χρόνια, σχετικά με τα revolving doors, μια ομάδα αποκάλυψε ότι ο πρώην εκτελεστικός διευθυντής της ΕΜΑ είχε ε, δημιουργήσει μια επιχείρηση συμβούλων όχι μετά αλλά δύο μήνες πριν την αποχώρησή του. Επιχείρηση η οποία ε, ε, προσπαθούσε να βελτιώσει τις αιτήσει αδειοδότησης. Στην εποχή είχα πολύ δουλέψει για αυτή την περίπτωση. Θα πρέπει η ΕΜΑ αλλά και η Επιτροπή ε, να λάβουν υπόψη αυτή την εμπειρία και να μας πούν πώς στο μέλλον θα εγγυηθούν μια καλή εφαρμογή του άρθρου 16 του καταστατικού των υπαλλήλων. Οι κανόνες υπάρχουν, το θέμα είναι η εφαρμογή τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο και εγώ, όπως και ο κύριος Παναγιωτόφ, ζητώ αναβολή της απαλογής μέχρι την τελική γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου σχετικά με την ΕΜΑ. Όσον αφορά την ΕΦΣΑ, κατάλαβα πολύ καλά ότι η αποφάσιση του διαμεσολαβητή της 7ης Δεκεμβρίου ε, προκάλεσε αντίδραση, αλλά εδώ και δύο χρόνια έχουμε επιτάπητο στο θέμα αυτό, το οποίο πρότεινα εγώ και άλλοι ευρωβουλευτές, όπως κυρία Σουντρένκενς, πρώην συντονίστρια επιστημονική και επικεφαλής της μονάδας για τα μεταλλιγμένα ε, προϊόντα, ο διαμεσολαβητής έκανε τρεις συστάσεις ε, να ενισχύσουμε τους κανόνες για την θέση των υπαλλήλων που θα πρέπει να αποκαλύψουν τα στοιχεία τους. Η ΕΦΣΑ, η ΕΑΑΤΑΦΑ, ΕΕ, δεν είδε τις δυνατότητες συγκρούσεως συμφερόντων. Εάν κάποιος παρουσιαστεί και πάλι, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων να έχει μια καλή ε, περιγραφή ε, των, ε, των λειτουργιών, των εργασιών για να δούμε αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Δεύτερον, από μια άποψη πιο γενική. Από το 2010 η επανάληψη συγκρούσεως συμφερόντων σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα μεταλλαγμένα προϊόντα και την υπόθεση της ασπαρτάμης που είναι κάτι που δεν είναι φυσικό. Παραλήψεις αναφοράς της δήλωση σύγκρουση συμφερόντων νομίζω θίγει την αξιοπιστία του της αρχής ενώ χρειαζόμαστε αυτόν τον οργανισμό και μιας πραγματογνωμοσύνης την οποία θα πρέπει να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Το Pesticide Net Action Network είδε, έλεγξε από απόψεως τοξικολογίας, την εργασία της ΕΦΣΑ και τις σχέσεις με τον βιομηχανικό κλάδο. Αυτή η σύγκρουση συμφερόντων αφορά επίσης και τα μεταλλαγμένα προϊόντα, το Requiter, από την και ένα πάνελ είχε συνεργαστεί με την βιομηχανία για τις μεθόδους αξιολόγησης των κινδύνων σε διάφορα φόρουμ, όπως η ύψη. Η ύψη επηρέασε τις ε, κατευθυντήριες γραμμές ε, για τα μεταλλαγμένα προϊόντα και νομίζω ότι γι' αυτό θα μιλήσουμε αργότερα. Το 2006 ο Γκλέν από την Monsanto, επικεφαλής μιας ε, task force, σε ένα συμπόσιο στην Αθήνα, είδε μεγάλον αντίκτυπο πάνω στις κατευθυντήριες γραμμές. Αυτό δεν είναι φυσικό. Ζητούμε λοιπόν μια συζήτηση για την σκοπιμότητα για την ΕΦΣΑ να ενημερώνει τους εμπειρογνώμονες των σχέσεων που θα πρέπει να έχουν με την ήλση. Τα 15 βιομηχανικά μέλη της ήλση που παράγουν τρόφιμα, χημικά προϊόντα και φαρμακευτικά προϊόντα. Είναι σημαντικός ο όμιλος αυτός. Το θέμα αυτό επανέρχεται συνεχώς ε, και το έργο της Ήλση ε, έχει κατακριθεί από το Μαγκόσμιο Οργανισμό Υγείας λόγω των σχέσεων με ε, την καπνοβιομηχανία. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για την επίλυση όλων των προβλημάτων. Η Ευρωπαϊκή Αρχή προσπαθεί να λάβει υπόψη τον ορισμό του όσα, αλλά τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εντάσσουν έναν ακριβή ορισμή του τι εννοεί η ΕΦΣΑ με συγκρούσεις συμφερόντων κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 16 του καταστατικού των υπαλλήλων, ένα σύστημα διασταυρούμενης επαλήθευσης με τα στοιχεία της βιομηχανίας και τον προσδιορισμό ε, κυρώσεων σε περίπτωση εκούσιας παράληψης ε, στις ε, δηλώσεις. όταν, όταν, εφόσον δεν έχουμε απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, θα πρέπει να ζητήσουμε μια αναβολή. Με συγχωρείτε που μακρηγόρησα, αλλά είναι σημαντικό το θέμα και τώρα δίνω τον λόγο ε, στον κύριο Ζερπόντι, τον συνάδελφό μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και να σας ευχαριστήσω και για τα όσα είπατε εσείς. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τη Γιούτα Χάουκ που λέει ότι είναι ελάχιστοι οι συνάδελφοι που είναι παρόντες ε, όταν συζητούμε τα θέματα της απαλλαγής. Να σας υπενθυμίσω ότι η Όλκα Πόνε φυλακίστηκε διότι έληξαν τα φορολογικά του βιβλία και είδαν ότι δεν είναι εντάξει και αυτό ήταν ο μόνος τρόπος για να μπει στη φυλακή. Νομίζω ότι είναι το μόνο λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε εμεί ω Επιτροπή για την προστασία του περιβάλλοντος ε, η απαλλαγή. Και έχω και μια ερώτηση από αυτού. Συμφωνώ πολύ με το σχέδιο γνωμοδότησης της κυρίας Χάουγκ και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο λόγος να τα αλλάξουμε όσα λέει, αλλά η ερώτησή μου είναι για τους άλλους τομείς πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε περιορισμένοι μόνο σε θέματα περιβάλλοντος ή ως ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος μπορούμε να σχολιάσουμε και την κοινή γεωργική πολιτική και την κοινή αλληλευτική πολιτική. Και το ρωτώ αυτό διότι ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού έχω το προνόμιο να λαμβάνω πολλές εκθέσεις από το ελεγκτικό συνέδριο και είναι πάρα πολύ επικριτική Ιδίω ε, για τα περιβαλλοντικά στοιχεία σε άλλα προγράμματα. Για παράδειγμα, ε, το πρόγραμμα περιβάλλοντος ε, γεωργίας στην ΚΑΠ εμείς επιτυγχάνουμε μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των περιβαλλοντικών στόχων αυτού του προγράμματος που είναι στοχευμένο προς το περιβάλλον. Ω Επιτροπή λοιπόν μπορούμε να είμαστε πολύ επικριτικοί επί του θέματος. Επιπλέον, την περασμένη εβδομάδα το Ελεγκτικό Συνέδριο έκανε μια έκθεση για την ε, κοινή αλληλευτική πολιτική. Τη δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα και ε, επιτέθηκε σε θέματα της υπεραλίευση. και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν καθορίζεται καν η δυνατότητα του αλληλευτικού στόλου. Ε, στο, στην κοινή αλληλευτική πολιτική. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι εάν μπορεί η Επιτροπή Περιβάλλοντος να ασχοληθεί και με τα άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαι διατεθειμένος, παρά το γεγονός ότι αύριο είναι η προθεσμία, ε, να καταθέσω και τροπολογίες από αυτόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Ριπαζή. Ε, merci, ε, merci Madame la Présidente. Je suis vraiment tout à fait d'accord avec votre intervention. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και την παρέμβασή σας για την ΕΦΣΑ και την Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων. Και ευχαριστώ και την κυρία Χαούκ για όσα είπε για τον προπολογισμό. Ξέρω ότι αυτό που θα πω δεν είναι η άποψη πολλών, αλλά ορισμένες ε, ε, Εταιρείε όπω η να χρηματοδοτείται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από τα τέλη των εταιριών ε, των φαρμακευτικών που θέλουν να περάσουν τα φάρμακα στην ε, αγορά. Αυτό δεν μου φαίνεται ότι είναι καλό, γιατί αν υπάρχουν πολλά στις φορές από τη βιομηχανία, ε, συχνά δημιουργούνται κάποιες παφέ που διευκολύνουν τη σύγκρουση συμφερόντων. Όσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίε, εκπλήττομαι. Ένας έλεγχος που έγινε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων από υπαλλήλου τη Επιτροπής χρειάστηκαν ε, δύο χρόνια σε μια ένωση, την Formindep Γιατρών, ε, για να την έχουν και ζήτησαν από τον διαμεσολαβητή να έχουν πρόσβαση σε αυτό το έγγραφο που είναι ένα δημόσιο έγγραφο. Ήδη υπάρχει μια δυσλειτουργία. Πώς συμβαίνει, ενώσεις, οργανώσεις, ε, και εμεί, μέλη του Κοινοβουλίου να μην έχουμε πρόσβαση σε αυτού του εσωτερικού ελέγχου, που είναι ο έλεγχο τη 30 η Απριλίου 2009 έχουμε ένα δεύτερο έλεγχο του 2010 γιατί δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτόν τον έλεγχο διότι αν θέλουμε να δούμε την εξέλιξη που ζητούμε για τι συγκρούσει συμφερόντων για την διαχείριση αυτών των οργανισμών θα πρέπει να μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα αυτών των εσωτερικών ελέγχων δεύτερο για τη σύγκρουση συμφερόντων με έκπληξη έμαθα και ξέρετε ότι ο Λόγκρεν είχε κατακριθεί όταν μάθαμε ότι ήταν ε, μέλος ενός γραφείου συμβούλων, αλλά το γεγονός ότι μάθαμε ότι ήδη τον Νοέμβριο, το Νοέμβριο είχε ήδη το δικό του γραφείο, ενώ έφυγε δύο μήνες μετά, αποχώρησε δύο μήνες μετά. Αυτή είναι μια λύση λειτουργίας από διαρθρωτικής πλευράς. Και τι ε, μαθαίνουμε, ότι έλαβε ένα εκατομμύρια δολάρια από την φαρμακοβιομηχανία υπομορφή stock options μετοχών, ε, διότι ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένες ε, οι φαρμακοβιομηχανίες. Δεν μπορούμε να έχουμε ε, σε σχέση με το διορισμό του κάτι το αναδρομικό, διότι αυτό είναι αντίθετο με το άρθρο 16 που αναφέρεται κυρία Πρόεδρε και αυτό από συμβολικής απόψεως θα ήταν αρκετά δυνατό να πούμε ότι δεν δικαιούστε να είστε μέλος ενογραφείου συμβούλων για να συμβουλεύετε ε, τα εργαστήρια των φαρμακοβιομηχανιών για να μπουν ορισμένα φάρμακα στην αγορά. Ε, σε αυτόν τον έλεγχο τι μαθαίνουμε, ότι οκτώ φάρμακα ε, αδειοδοτήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, με εμπειρογνώμενος, οι οποίοι ήταν κριτές και ενδιαφερόμενοι. Δηλαδή, τους αναθέτουμε εκθέσεις για ένα φάρμακο και έχουν μετοχές στην φαρμακοβιομηχανία που θα παράγει αυτό το φάρμακο μετά τον έλεγχο έγινε επαναξιολόγηση αυτών των οκτώ φαρμάκων, διότι αν αδειοδοτήθηκαν μετά πραγματογνωμοσύνη εμπειρογνωμόνων που ήταν μέλη εργαστηρίων ε, φαρμάκων, εμείς δεν έχουμε καμία εγγύηση ότι τα φάρμακα αυτά δεν έχουν παρενέργειες. Θα πρέπει να προσθέσουμε λοιπόν πολλά πράγματα σχετικά με την λειτουργία των οργανισμών, σχετικά με την αρχή ασφάλειας τροφίμων. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Λεπάζ και νομίζω ότι ένα από τα στοιχεία για να ενισχύσουμε το ρόλο των Ευρωβουλευτών είναι να μην ψηφίσουμε αυτή την απαλλαγή, διότι αν την ψηφίσουμε θα συνεχίσουν. Ζητούμε να υπάρχουν άμεμπτες ε, οργανώσεις ευρωπαϊκές τα εργαστήρια λένε ότι είναι πιο εύκολο να λάβουν μια άδεια για την εμπορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο από ότι σε εθνικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Αν είναι πιο εύκολο να πουλούνται στην Ευρώπη, αυτή η αγορά είναι πολύ μεγαλύτερη από την εθνική, από κάθε εθνική αγορά. Εγώ λοιπόν επιβεβαιώνω και ενισχύω, ε, υποστηρίζω την ιδέα της Πρόεδρου Λοπάς και θα ήθελα και η συγγήτρια να ακολουθήσει αυτή τη γραμμή για να δώσουμε το παράδειγμα ότι θέλουμε οργανισμούς και αρχές που να είναι αμέμπτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ κυρία Λιμπεζία. Η κυρία Ζόφια Μαζέκ Μπουκοβίτς. καταρχήν πρέπει να για την τόσο αναλυτική έκθεση. Δεν να μου πείτε κάτι περισσότερο. Πώς αντιδράσαν οι υπηρεσίες αυτές στην σημερινή οικονομική κρίση, Κατά πόσο προσανατολίστηκαν στην ε, κρίση αυτή σε κάποιους γιατί βέβαια ξέρουμε ότι το θέμα της υγείας εξαρτάται από το περιβάλλον, από την διατροφή, αλλά και το πώ αισθάνεται κανεί. Κάποιο δηλαδή που κάνει την θέση εργασία του έχει πιο πολλά ε, προβλήματα υγεία. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω για τι υπηρεσίε τι κάναν προ την κατεύθυνση αυτή. και την κατανόηση των ε, πολιτών. Γιατί ξέρουμε σήμερα ότι και ε, τα μία περίθαλψης ε, μειώνουν, ε, στα ταμεία περίθαλψης μειώνεται το αποθεματικό συνεχώς, λόγω ακριβώς της κατάστασης του, της ίδιας του πληθυσμού. Και θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη κατανόηση της υγιούς ζωής. Η κυρία Όκεν. Θα είμαι πολύ σύντομη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να υποστηρίξω και αυτό που είπατε και εσείς, κυρία Πρόεδρε διότι ασχολούμαστε με τόσα πολλά προβλήματα για κάποιες από αυτές τις υπηρεσίες και θα ήθελα να δω και τις ε, σχέσεις που ισχύουν η αίμα πλέον είναι υποχρεωμένη να ε, έχει μια κάποια διαφάνεια. Υπήρχε πόλεμος στην αρχή. Γνωρίζω από το Σκανδιναβικό Ινστιτούτο ότι υπήρχε πόλεμος. Το περασμένο καλοκαίρι υπήρχε διαμάχη, πολύ μεγάλη επί του θέματος. Είναι πολύ κλειστά όμω τα συστήματα. Γνωρίζω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο κάποιοι δεν μπορούν καν να λάβουν πληροφορίε ε, για πηγέ κλινικών δοκιμών, ακόμα και αν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά και δείχνουν ε, ε, επικίνδυνα στοιχεία. Τα κρατούν ω στο μυστικό και αυτό είναι σχεδόν εγκληματικό. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να δούμε τι κάνουμε με αυτού του τόσο σημαντικού οργανισμού και τη σχέση μεταξύ των εθνικών αντίστοιχων οργανισμών και των ευρωπαϊκών οργανισμών. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός παραδέχτηκε πλέον ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Αλλά δεν ισχύει αυτή τη στιγμή. Και αφού είναι τόσο αλληλένδετα όλα αυτά, ε, είναι απαραίτητο να είμαστε αυστηροί και να ακολουθήσουμε σκληρή γραμμή, διότι εμείς πρέπει να προστατεύσουμε την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Ναι, συμφωνώ πλήρως μαζί σας, η κυρία Τεστόρη για την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ, κυρία Διευθύντρια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ε, λαμβάνω τον λόγο ε, ξέρω ότι δεν πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά απλώ θα ήθελα να σας πω πόσο ο Επίτροπός μου αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις συγκρούσεις συμφερόντων. Και εδώ και εννέα μήνες έχουμε μια ε, ειδική ομάδα με όλους τους οργανισμούς ε, για να είμαστε βέβαιοι ότι η CDC, η ΕΜΑ, η ΕΦΣΑ να εφαρμόζουν τα πρότυπα, τους κανόνες, τους πιο αυστηρούς για τις συγκρούσεις συμφερόντων, για τις περιπτώσεις για τις οποίες μιλήσατε για τις περιπτώσεις που μας ανησυχούν, αλλά είναι περιπτώσεις του παρελθόντος. Τώρα έχουμε θεσπίσει μια πολιτική για τις συγκρούσεις συμφερόντων στους οργανισμούς που είναι η πιο αυστηρή δυνατή και μπορούμε να σας παρουσιάσουμε τις λεπτομέρειες όποτε θέλετε κυρία Πρόεδρε και εξάλλου σκεφτόμαστε να εκπονήσουμε μια έκθεση που θα παρουσιάσουμε στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο για το τι έκανε η DG Sanko από τότε που ανέλαβε αρμοδιότητα για την αίμα, για τα φάρμακα και την ΕΦΣΑ για την ασφάλεια τροφίμων. Ευχαριστώ κυρία Διευθύντρια. Μήπως θέλετε να λάβετε το λόγο κυρία Ισηγήτρια. Ναι, καταρχήν έχω μία παράκληση. Και εσείς κύριε Λεπάς και Μουσέλ Ριβαζή και η κυρία Όκαν συμφώνησα με αυτό που είπατε εσείς. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα, μια που το έχετε γραπτά αυτά που είπατε, να μου το δίνατε και εμένα γραπτά. Πρώτα αυτό, πολύ ωραία. Δεύτερον, κάποιος ρώτησε κατά πόσον εμείς ως Επιτροπή Περιβάλλοντος έχουμε να πούμε κάτι και σε άλλους τομείς πολιτικής κατά τη διάρκεια της Όχι. Θα πρέπει να πάμε στις άλλες επιτροπές και αυτό εννοούσα. Ξέρω. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος Ό,τι συζητάμε τώρα τη μεταρρύθμιση είναι θέμα της, Επιτροπής Πολιτικ... της Πολιτικής ε, Συνοχής, ε, Γεωργίας, ε, Αλίας κλπ. Εμείς πρέπει να γνωμοδοτήσουμε αλλά μας ξέρω, να το πω έτσι. Αφήνουμε τον εισηγητή να προετοιμάσει την ε, γνωμοδότηση, Ενδεχομένω κάνουμε και κάποια τροπολογία από αυτές Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι να ασχοληθούμε πραγματικά άμεσα με τις προτάσεις κομισιών Κομισιόν ως βουλευτές και να συζητήσουμε τους συναδέλφους μας στις πολιτικές μας ομάδες για να δούμε ποια θα πρέπει να είναι η κατεύθυνση της μεταρρύθμισης. Αλλιώ δεν πρόκειται να καταλήξουμε σε, σε αποτέλεσμα. Έτσι κι αλλιώς όλα είναι αλληλένδετα. Ελπίζω όμω να μπορέσουμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό που είπε Πάολο Τσεστόρη μόλι τώρα είναι σωστό. Ασχολούμαστε με το παρελθόν. Το έτος 2010. Έτσι έχουν τα πράγματα όταν ασχολείται κανένας με την απαλλαγή. ολοκληρωμένο προπολογισμό ενό έτου είναι η αφορμή για να ασχοληθούμε με αυτό. Είναι σαφέ. Το πρόβλημά μου είναι πρόβλημα πολλών. Αλλά και το πρόβλημα ας πούμε της Μίσελ Ριβαζή που λέει ότι εγώ θέλω να δω τους εσωτερικούς ελέγχους. Να έχω όλα τα στοιχεία ανοιχτά στα χέρια μου. Αγαπητοί συναδελφοί, αυτή η εσωτερική έλεγχη όπως είναι άσχετα αν πρόκειται για υπηρεσίες ή αν πρόκειται για τμήματα της Κομισιόν που εσωτερικά ελέγχονται. Εσωτερικοί αυτοί έλεγχη έχουν σαν στόχο να μπορούν να υπάρχουν διοικητικές νομοθετήσεις, τοποθετήσεις και βελτίωση ενδεχομένως κάποιες κατάστασεις. Καταλαβαίνετε ποια μορφή θα έχουν αυτοί οι εσωτερικοί έλεγχοι εάν ε, προσεχώς θα πρέπει να είναι στην ε, ιστοσελίδα. Ε, εάν εγώ είμαι ένας από τους θα εκθέσω τους συναδέλφους και θα λέω δημόσια αυτό και αυτό και αυτό ε, το κάνατε στραβά και θα πρέπει να το κάνετε διαφορετικά. Γι' αυτό λέγονται εσωτερικές, ε, εσωτερική έλεγχη αυτή για να μην εκτίθεται κανένας και να μπορεί όμως να ακουστεί αυτό που είναι απόλυτα στραβό. Μέσα στα πλαίσια της απαλλαγής, ο εισηγητής έχουν τη δυνατότητα να ρίξει μια ματιά σε αυτούς τους ελέγχους για να τους λάβει υπόψη και εγώ δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ μαζί σας. Δεν συμφωνώ με τον διαμεσολαβητή. Ότι κάποιος τυχαίος δημοσιογράφος που θέλει να, ε, να εκφραστεί κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορεί να έχει εσωτερικούς ελέγχους στα χέρια του. Απαγορεύεται αυτό. Δεν επιτρέπεται εμείς ως βουλευτές μπορούμε μεμονωμένα να εξετάσουμε αυτούς τους ελέγχους αλλά δεν υπάρχουν στην ιστοσελίδα. Αυτή είναι η δική μου πεποίθηση 100% γιατί ε, πιστεύω ότι αν αυτή η εσωτερική ενοχή, όχι η λογιστική ενοχή που έχει το ηλεκτρικό συνέδριο, αυτό είναι για όλους και σωστά. Αλλά αν η εσωτερική αυτή η διατίθενται δεν θα πέτυχαν το στόχο τους γιατί θα πρέπει να βοηθήσουν τη βελτίωση της διοίκησης. Και αν είναι δημόσιοι δεν θα έχουν πια κανένα νόημα. Καταλαβαίνω, διαφάνεια, διαφάνεια, εντάξει. Είμαι υπέρ της διαφάνειας, αλλά η διαφάνεια θα πρέπει να είναι σωστή. Η διαφάνεια σημαίνει ανοίγουμε τα πάντα. Αλλά τώρα δεν θα χρειάζεται αυτή η μονάδα των εσωτερικών ελέγχων. Τι θα κάνουνε. Τι θα κάνουνε. Και στο εσωτερικό του κοινοβουλίου υπάρχει κάτι τέτοιο. εσωτερική ελεγχτές. Που λένε, για κοιτάξτε εδώ, αυτό δεν πάει καλά, κάντε αυτό αλλιώς και βελτιώστε τη στάση σας εκεί. Σωστό αυτό, πολύ καλό. Αλλά όλα αυτά είναι ανοιχτά, ώστε ο καθένας να μπορεί να με φτύνει, ας πούμε, αν κάτι δεν έχει, έχω κάνει καλά, το μόνο που καταφέρνω δεν είναι να έχω περισσότερη διαφάνεια, αλλά να αποτρέπω την καλή εργασία. Qu'on passe au sujet suivant, Michel. Euh, oui, très, très rapide, mais c'est essentiel la discussion que l'on a. C'est jusqu'où on ouvre. Ναι, θα ήθελα να πω μέχρι που μπορούμε ε, να διαβιβάζουμε τα αποτελέσματα σε όλο το κοινό. Εμένα μου φαίνεται και αναφέρομαι σε αυτά που συμβαίνουν ε, με την Food and Drug Authority στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα είναι διαφανή, όλα είναι προσβάσιμα στο διαδίκτυο. Ε, έχουμε το, τον εσωτερικό έλεγχο. Ο εσωτερικό έλεγχο επιτρέπει να δούμε την λειτουργία και εφόσον γίνονται έλεγχοι κάθε χρόνο μπορούμε να δούμε ε, πώς βελτιώνονται οι κριτικές με τον εσωτερικό έλεγχο. Δεν είμαστε εδώ για να διαλύσουμε οργανισμούς. Χρειαζόμαστε τους οργανισμούς αυτούς. Πρέπει να τους βελτιώσουμε. Και για να τους βελτιώσουμε πρέπει να έχουμε πρόσβαση στα έγγραφα. Και ο ρόλος της Επιτροπής για την οποία μιλήσατε είναι ακριβώς να κάνει απολογισμό όλων αυτών των ελέγχων. Πρέπει να γίνει σημαντική εργασία ανάμεσα στο ελεγκτικό συνέδριο, μεταξύ των εξωτερικών ελέγχων κλπ. Πρέπει να έχουμε τα ε, έγγραφα όμως που να είναι διαθέσιμα, αλλά όχι εμπιστευτικά με τις πληροφορίες. Και όταν, και όταν μιλάμε για διαφάνεια, ε, πρέπει να έχουμε διαφάνεια. Ακόμα και οι επιτροπές που θα δώσουν τη γνωμοδότησή τους για ένα φάρμακο, έχουμε το θέμα της υπευθυνότητα. Θα πρέπει ένας εμπειρογνώμονας να δώσει επιχειρήματα γιατί επιτρέπει ή δεν επιτρέπει ένα φάρμακο. Εάν έχουμε μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων, των οποίων δεν ξέρουμε τα ονόματα, δεν ξέρουμε ποιο αποφασίζει τι, ε, εκεί έχουμε συγκρούσεις συμφερόντων σημαντικές, διότι πιστεύουν ότι προστατεύονται τη μη διαφάνεια. Εγώ νομίζω ότι η διαφάνεια πρέπει να είναι Όλα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Η Πρόεδρος, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε βεβαίως πέραν από τον προϋπολογισμό και θα ήταν καλό να οργανώσουμε μια συζήτηση με κάποια μορφή στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2012. Αυτά είναι θέματα τα οποία είναι μείζονος σημασίας. Ναι, ναι. Ο κύριος Σίμπερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δυστυχώ ο δικό μα σκιώδη συζητητή δεν είναι εδώ. Γι' αυτό παίρνω εγώ το λόγο και θα ήθελα ρητά να υποστηρίξω τα επιχειρήματα τη συναδελφού ε, Χάουκ. Γιατί εδώ δεν θέλουμε με τη διαδικασία αυτή απαλλαγή να δημιουργήσουμε μία απλή διαφάνεια, αλλά θέλουμε οι ευρωπαϊκέ αυτέ υπηρεσίε να λειτουργούν και προ όφελο των πολιτών γιατί εσωτερικές εκθέσεις, εσωτερικές έλεγχοι, αν έχουν νόημα θα πρέπει εμείς ως βουλευτές να μπορούμε να τις ε, διαβάζουμε τους αποτελέσματα αυτά για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Αλλά αν περάσει στην ιστοσελίδα τότε πραγματικά θα έχουν πολύ νόημα. Πολλές από τις εκθέσεις αυτές σχετίζονται και με την πνευματική ιδιοκτησία όσον αφορά αυτές τις διαδικασίες ελέγχου. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει αρκετή ε, αντικειμενικότητα, αλλά δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε άμεσα κανέναν. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό στη διαδικασία αυτή απαλλαγής να ε, δείξουμε πόσο αποτελεσματικοί είμαστε στην προσπάθεια επιτυχίας καλής λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών. Και οπωσδήποτε, όπως είπατε και εσείς, ε, το θέμα των υπαλλήλων που αλλάζουν από τη μια στην άλλη θα πρέπει να δούμε μήπως ο κώδικας συμπεριφοράς είναι κάτι που θα πρέπει να εισαγάγουμε. γιατί πραγματικά η υπερβολική διαφάνεια στα εσωτερικά θέματα δεν θα βοηθήσει, θα είναι μάλλον αρνητική επί Και ευχαριστώ για άλλη μια φορά την Γιούτα Χαόκ που νομίζω ότι εργάστηκε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ άλλη μια φορά. Ευχαριστώ την κυρία εισηγήτρια για την σημαντική αυτή εργασία. Υπενθυμίζω πως τονίσατε ότι η κατάθεση τροπολογιών είναι ε, στις 20 ε, ε, Δεκεμβρίου στις 18 η γενική ψηφοφορία το Μάρτιο. Και τώρα περνάμε στο σημείο 16, 16, 13 με συγχωρείτε τη ημερήσια διάταξη σχετικά με την έκθεση αξιολόγηση τη νομοθεσία για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Κυρία Διευθύντρια, αν έχετε την καλοσύνη να λάβετε το λόγο και να μας πείτε περί τίνος πρόκειται. Ευχαριστώ, πολύ και σας ευχαριστώ πολύ διότι μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω την αξιολόγηση της νομοθεσίας για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς την οποία ολοκληρώσαμε το περασμένο φθινόπωρο. Η αξιολόγηση αυτή είναι στμήμα της συνεχούς διαδικασίας που εφαρμόζουμε στην νομοθεσία μας για να αξιολογούμε συνεχώς εάν είναι η κατάλληλη νομοθεσία βάσει των προκλήσεων που αντιμετωπίσουμε. Στον τομέα των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών θα ήθελα καταρχάς να σας παρουσιάσω κάποια στοιχεία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο γενετικώς ε, τροποποιημένοι οργανισμοί που ε, χρησιμοποιούνται. Η ε, Monsanto 811 που είναι αραβόστο που καλλιεργείται σε πέντε κράτη-μέλη και αμφλόρα πατάτα η οποία καλλιεργείται σε τρία κράτη-μέλη. Αυτά είναι τα δύο γενετικώς τροποποιημένα είδη που καλλιεργούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή έξι κράτη-μέλη τα οποία έχουν ε, λάβει ρήτρα ασφαλεία ε, κατά ε, ενό ή και των δύο αυτών των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών. Σήμερα δεν υπάρχει καμία επισήμανση για γενετικό τροποποιημένο οργανισμό ε, στην αγορά, ε, σχεδόν καμία επισήμανση, διότι αν, πρέπει να, ε, αν περιλαμβάνει γενετικό τροποποιημένος οργανισμός πρέπει να επισημάνονται. Υπάρχουν κάποια φασόλια σόγιας και μαγιονέζα που εισάγονται. Αντίθετα, όσον αφορά τις ζωοτροφές, το 85 με 95% των ζωοτροφών στην αγορά είναι προέλευση γενετικώ τροποποιημένων οργανισμών και υπάρχει ανάλογη επισήμανση. Οι δύο αξιολογήσει που εξετάζουν ε, την περιβαλλοντική νομοθεσία και την νομοθεσία για, τις, ε, για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές ε, και τους γάματα φαόμικρων καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η απάτη δεν απορρέει από την ίδια την νομοθεσία αλλά από την εφαρμογή της η οποία γίνεται σε ένα πολύ δύσκολο πλαίσιο σε διεθνές επίπεδο και είναι και ανισόρροπη σε επίπεδο κρατών μελών. Οι δύο εκθέσεις λοιπόν καταδεικνύουν ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερη εφαρμογή και ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα μέτρα για πιο εναρμονισμένη εφαρμογή. Θα συνοψίσω τώρα ποια είναι οι διαπιστώσεις των αξιολογήσεων αυτών. Καταρχάς, οι αξιολογήσεις λένε ότι χρειαζόμαστε περισσότερες ρητές κατευθυντήριες γραμμές ε, αξιολόγησης κινδύνου που θα υιοθετηθούν από όσου ε, εξετάζουν τα θέματα κινδύνου ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι κατά την αξιολόγηση κινδύνου θα γίνεται ε, μια αξιολόγηση που θα βασίζεται σε συγκεκριμένες κατευθυντήρες γραμμές. Δεύτερον, η αξιολογή για του γενετικώ τροποποιημένου οργανισμού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται περισσότερη ευελιξία στα κρατημέλη και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντε. Τρίτον, όσον αφορά τα εισαγόμενα προϊόντα, η αξιολόγηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας έγκρισης και επίσης να αντιμετωπίσουμε και τα περιστατικά χαμηλής παρουσίας, τα LLP, στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω ε, διαφορετικής ταχύτητας κατά την έγκριση εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών, η αξιολόγηση καταλήγει ότι καλύτερο θα ήταν να έχουμε μια εθελοντική προσέγγιση, αλλά πρέπει να υπάρχει μια προσέγγιση που θα ε, αναπτυχθεί βάσει εναρμονισμένου πλαισίου. Θα ήθελα να καθησυχάσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Έχουμε λάβει πολύ σοβαρά υπόψη την αξιολόγηση και έχουν εφαρμοστεί ήδη κάποια μέτρα για να απαντήσουμε στα όσα προκύπτουν από την αξιολόγηση. Και θα ήθελα να σας παρουσιάσω συνοπτικά αυτές τις δράσεις. Ως προς την καλλιέργεια, καταρχάς έχουμε εγκρίνει το πακέτο καλλιέργειας για το οποίο έχει ήδη γνωμοδοτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτά συζητώνται αυτή τη στιγμή και στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεύτερον, για θέματα παρουσίας ε, σε χαμηλό ποσοστό έχουμε, εφαρμόσει, έχουμε εγκρίνει εφαρμοστικούς κανόνες οι οποίοι προσπαθούν να έχουν μια εναρμονισμένη προσέγγιση για τον έλεγχο της χαμηλής παρουσίας γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και αυτά εφαρμόζονται από τον, ε, από τον Ιούλιο του 2011. Τρίτον, για τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δημοσίευσε τον Απρίλιο μία έκθεση για αυτές τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις των καλλιεργών ε, γεωνετικώς τροποποιημένων οργανισμών βάσει των στοιχείων που λάβαμε από τα κράτη-μέλη και ξεκίνησε και μια διαδικασία βάσει τη οποίε έγινε και μια σημαντική διάσκεψη στην οποία συμμετείχαν και ευρωβουλευτές ε, τον Οκτώβριο. Για την αξιολόγηση κινδύνου τώρα, ε, ολοκληρώνονται οι κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση κινδύνου για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και όπως είπε και ο Επίτροπος ε, θα αποσταλεί σχέδιο κειμένου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζουμε να μπορέσουμε να εγκρίνουμε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές στις αρχές ε, του επομένου έτους και επίσης αναθεωρούμε επίσης και τι κατευθυντήριε γραμμές για την ε, αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για την επισήμανση τώρα των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών ξεκινά μια μελέτη για να δούμε πώς θα μπορούσαμε να έχουμε ένα αρμονισμένο σύστημα και κατά πόσον χρειαζόμαστε ένα αναρμονισμένο σύστημα. Και τέλος, όσον αφορά την παρακολούθηση, διότι ο Επίτροπος επιμένει ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί και η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συζητούμε αυτή τη στιγμή με τα κρατη και τις αρμόδιες επιχειρήσεις για να δούμε εάν μπορούμε να έχουμε πιο εμπεριστατωμένες κατευθυντήρες γραμμές, ώστε να έχουμε αποτελεσματική ε, περιβαλλοντική παρακολούθηση μετά από την έγκριση και οργανώνεται για τον επόμενο Μάρτιο και σχετική ε, διάσκεψη. Νομίζω λοιπόν, κατακλείδη, ότι είμαστε στο σωστό δρόμο, αλλά χρειαζόμαστε και προσπάθεια από όλες τις πλευρές, ιδίω από τα κράτη-μέλη, ώστε να βεβαιωθούμε ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας μας θα ε, συνεχίσει να γίνεται με αποτελεσματικό και εναρμανισμένο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, Ευχαριστώ κυρία Διευθύντρια. Κυρία Μακάβαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επιτροπή για αυτήν την παρουσίαση. Χαιρετίζω το τελευταίο σημείο που αναφέρεται σχετικά με την περιβαλλοντική αξιολόγηση, διότι μας ενδιαφέρει πολύ ο αντίκτυπος πάνω στην βιοπικιλότητα. Είχαμε ε, εκθέσεις ε, για προβλήματα στην Ινδία. Όχι μόνο αντίκτυπος στις καλλιέργειες, αλλά και για μετατόπιση. Και θα ήθελα η Κομισιόν να εξετάσει αυτά τα πράγματα πού έχετε μια καλλιέργεια ε, παραμπτός χάρη βάμβακος και τα έντομα τα οποία ανθίστανται και μεταναστεύουν σε καλλιέργειες τροφίμων και καταστρέφονται ε, για τον τοπικό πληθυσμό. Ε, διότι αυτές είναι οι καλλιέργειες που προσελκύουν τα έντομα. Αυτά θα πρέπει να, ε, να εξετάσουμε, διότι ε, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν ξέρω αν θα έχω επιπτώσεις αν φάω γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, αλλά πρέπει να εξετάσουμε και αυτά τα προβλήματα και να έχουμε τα αποτελέσματα εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, Λίντα Μακαβάν. Ο κύριος Βάντελεν. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Βλέπω ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή επιμένουν στο ρόλο το οποίο έχουμε κληθεί να παίξουμε και έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα για το 2012. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα ε, στην ε, κυρία Διευθύντρια σε σχέση με μια έκθεση που εκπονήθηκε από μια ομάδα εργασίας ε, για τις νέες τεχνικές. Υπάρχουν ορισμένες τεχνικές που αποτέλεσαν αντικείμενο εξέτασης και ανάλυσης και θα ήθελα να επιμείνω πάνω στο γεγονός ότι έχουμε ε, μια ημερομηνία για μια έκθεση που είναι ο Μάρτιος 2011 ε, ε, σχετικά με τις νέες τεχνικές που μελετήθηκαν ελπίζω να έχουμε τα αποτελέσματα της έκθεσης αυτής αρκετά γρήγορα διότι εδώ και ένα χρόνο περιμένουμε για την δημοσίευση ορισμένων εκθέσεων την έκθεση της ΕΦΣΑ για την ασφάλεια ορισμένων προϊόντων και ορισμένων φυτών που έχουν τροποποιηθεί γενετικά, πότε μπορούμε να περιμένουμε αυτήν τη νέα έκθεση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Όκεν. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή τη, τώρα θα μιλήσω στα δανεικά. Θα έχω μερικές ερωτήσεις. τι συμβαίνει με τις μακροπρόθεσμες συνέπειες για το περιβάλλον. Τις λαμβάνουμε υπόψη ή όχι, διότι υπάρχει μια ολόκληρη σειρά διοδοτήσεων που συμπεριλαμβάνονται και εγώ θα ήθελα να μάθω μέχρι ποιου βαθμού λαμβάνουμε υπόψη τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Είδαμε τι συνέβη ε, με τις μέλισσες και αντιληφθήκαμε ότι δεν είχαμε λάβει υπόψη όλες τις επιπτώσεις. Αντιληφθήκαμε ότι υπήρχε πάρα πολύ μέλι που ήταν παράνομο διότι αυτό το μέλι δεν μπορεί να περιλαμβάνει ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Είχαμε σκεφτεί ότι θα μπορούσαμε να δούμε τι συνέβαινε με την αδειοδότηση, αλλά όχι, δεν λειτουργήσαν έτσι τα πράγματα και εδώ δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις μέλισσες, δεν ξέρουμε ε, πού θα πάνε, πού θα τραφούν από ε, διάφορα ε, λουλούδια που έχουν ψεκαστεί. Όχι, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις επιπτώσεις πάνω στο περιβάλλον. Εδώ δεν μπορούμε να λαμβάνουμε υπόψη μόνο τα οικονομικά στοιχεία και τα κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία. Έχετε όλες τις επιπτώσεις για τους παραγωγούς ε, μελιού, πράγματος. χάρη. Τι θα συμβεί τώρα, θα μπορέσουν να πουλήσουν αυτό το μέλι. Πώς θα μπορούμε ε, να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία μακροπρόθεσμα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα αυτά ε, τα στοιχεία μακροπρόθεσμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, η κυρία Χα προηγουμένως είπε ότι η διαφάνεια είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Θα έπρεπε η διαφάνεια να υπάρχει σε όλα τα επίπεδα πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ένα άνοιγμα ε, σημαντικό και ότι θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε όλα αυτά ε, με τα στοιχεία με τους εμπειρογνώμονες. Είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Και για να κλείσω, θα ήθελα να μάθω εάν θα μπορούσαμε να φανταστούμε πώς θα μπορούσαμε να υποχρεώσουμε κάποιους να τηρούν την Οδηγία 18 του 2001 παρά να βασίζομαστε στην Οδηγία του 2003 όταν πρόκειται ε, για τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα. Διότι εδώ έχετε ορισμένες διατάξεις που είναι πιο περιοριστικές Μπορεί να έχουμε ένα πρόβλημα υγείας, είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε πολύ καλά και αυτό θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις πάνω στην βιοπικιλότητα και από απόψεως ε, κοινωνικο-οικονομικής. Υπάρχουν θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που εμπλέκονται και θα μπορούσε να εκμηδενιστεί, να εξαλειφθεί κάθε φυσική καλλιέργεια. Ευχαριστώ. Η κυρία Σομέρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Κομισιόν για την έκθεσή τη. Εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις που πάνε πιο πέρα από αυτά που ακούσαμε. Δεν ξέρω αν μπορεί να απαντήσει η κυρία Στόλη. Αν θυμάμαι καλά, μας λείπουν ακόμα τα οριακά στοιχεία για, τα, ε, για τους πόρους προσφορά. Ξέρω ότι είναι μια άλλη γενική διεύθυνση, αλλά φαντάζομαι να επικοινωνείτε στην Κομισιόν. Έχετε συμπληρωματικές πληροφορίες μέχρι που έχουμε φτάσει. Και έχω και μια άλλη ερώτηση. γιατί φαίνεται ε, από τη συζήτηση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση κατα... υπάρχει μια εκτίμηση επιπτώσεων κατά πόσο θα ήταν δυνατόν στην Γεωργία να εργαστεί σήμερα κανένας χωρίς γενικά τροποποιημένους οργανισμούς συμπεριλαμβανομένων και των ζωοτροφών. Αν ξέρω καλά, εμείς εισαγάγουμε 70% των ε, ζωοτροφών πρωτεΐνες και τα περισσότερα από αυτά ε, από αυτές συμπεριλαμβάνουν ε, γεννητικά τροποποιημένους οργανισμούς. Υπάρχει δυνατότητα να αντικαταστήσουμε αυτούς τις ζωοτροφές με δική μας παραγωγή Ακούγεται αυτό, αλλά όπως το ξέρω δεν είναι δυνατόν και μόνο επειδή δεν έχουμε τις επιφάνειες και δεν έχουμε το σωστό κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν ξέρω, υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία από αυτόν. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ την Κορίνη που πρόεδρεσε και έχει το λόγο. Η ε, Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω κυρία Διευθύντρια μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τις ίδιες τις εκθέσεις. Υπάρχει μία η οποία ειλικρινά θα έπρεπε να αποτελέσει αντικείμενο μιας πραγματικής συζήτησης επί της ουσίας, διότι στόχος της νομοθεσίας. Δεν είναι να ευνοήσει την εμπορία των γενετικά μεταλλαγμένων οργανισμών. Είναι να προστατεύσει την υγεία και το περιβάλλον ε, στην, ε, κατά την διάθεση των οργανισμών αυτών. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έχουμε λοιπόν μια εκκίνηση, μια, αρχή, μια αρχική βάση η οποία είναι διαφορετική. Όταν τα κράτη-μέλη εκφέρουν αντιρρήσεις, το κάνουν για λόγους πολιτικούς και όχι για λόγους επιστημονικούς, λένε ορισμένες εκθέσεις. Δεν είναι σωστό αυτό. Υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη που βάσει των αξιολογήσεών τους έχουν ε, γνωμοδοτήσει επιστημονικά. Και τρίτον, νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα και έχουμε, το έχουμε ήδη συζητήσει, αναφέρεται στις συνθήκες εφαρμογής και συμμερίζομαι τα όσα είπε η κυρία Όκεν ε, πριν από λίγο η αξιολόγηση των αμέσων και μέσων κινδύνων, κυρίως ε, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Έχουμε την απόφαση του Συμβουλίου 2010, ε, έχουμε ε, την Οδηγία 18 για την βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και της ΕΦΣΑ. Συνεπώς εκπλήσωμε που έχουμε μια έκθεση που να έχει αυτήν την άποψη με τρόπο τόσο εμφανέ. Σημερίζουμε όμως το βασικό συμπέρασμα της Επιτροπής που λέει ότι δεν χρειάζεται να αναμορφωθεί η νομοθεσία για τους οργανισμούς αλλά να βελτιωθεί η εφαρμογή ο τρόπος της εφαρμογής αυτής της νομοθεσίας μπορεί να γίνουν προσαρμογέ σχετικά με την πρόταση για την καλλιέργεια είναι καλό πράγμα να, να επιτρέψει κανείς τα μελη να απαγορεύουν την καλλιέργεια και σε πρώτη ανάγνωση έχουμε ψηφίσει ένα κείμενο που ενισχύει την πρόταση της Κομισιό πρέπει να έχουμε μια αξιολόγηση του κινδύνου που να είναι λιγότερη στενή, λιγότερη στενή από αυτήν που έχουμε σήμερα, που να αναφέρεται σε όλες τις έμμεσες απόψεις και την σκοπιμότητα χρήσης των οργανισμών αυτών σε ένα αγρονομικό περιεχόμενο. Μας μίλησε η συνάδελφος για την Ινδία. Είναι σημαντικό και ενδιαφέρον να δούμε ε, πώς γίνονται τα πράγματα αλλού. Χαιρετίζω τις προσπάθειες της Επιτροπής για τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων. Υπάρχουν πρόοδοι κυρίως για τον αντίκτυπο των οργανισμών πάνω ε, στα έντομα που δεν είναι στόχοι. Πρέπει να δούμε την ισοδυναμία ως προς την ουσία που για μένα και για ορισμένους από εμά δεν είναι κάτι το αποδεκτό ε, όπου η συνεργατική αξιολόγηση των κινδύνων που απαλλάσσει τους οργανισμούς από κάθε διαδικασία. Έχω όμως μερικές διχογνωμίες για άλλα συμπεράσματα. Η σήμανση των προϊόντων που έχουν τραφεί με τροποποιημένους οργανισμούς. Υπάρχουν πάρα πολλοί παραγωγοί που, που τρέφουν τα πτηνά με, με οργανισμούς θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για αυτούς τους γεωργούς και κτηνοτρόφους να εξηγούν τον τρόπο που εργάζονται βλέπουμε την ιδέα ενός κατοφλιού ε, μετάδοσης ε, για τους ε, μη επιτρεπτούς οργανισμούς. Αν δεν επιτρέπονται, δεν επιτρέπονται. Γιατί να δεχθούμε ένα κατόφλι για κάτι που δεν είναι επιτρεπτό. Αυτό είναι αμφισβήτηση όλης της λογικής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής που βασίζεται στο σύστημα του τι επιτρέπεται και του τι δεν επιτρέπεται. Δεν μπορούμε να έχουμε κατόφλι για κάτι που απαγορεύεται και θέσπιση ενός κατοφλιού ε, μετάδοση στους σπόρους είναι ένα θέμα πάρα πολύ λεπτό και θα ήταν νομίζω παρανόηση κοινωνική, περιβαλλοντική, οικονομική. Θα μπορούσαμε να έχουμε οργανισμούς σε όλες τις απαρτίδες σπόρων χωρίς σήμανση. Και αυτό ανοίγει την πόρτα για μια ε, μετάδοση στην Ευρωπαϊκή Γεωργία με μια έκρηξη του κόστους για τον περιορισμό της μετάδοσης για αυτούς Πού θα το ήθελαν. Οι εταιρείε των σπόρων μπορούν να εξασφαλίσουν την καθαρότητα των σπόρων. Είναι πιο οικονομικό να ελαχιστοποιήσουμε την μετάδοση στα ανάντη, στην πηγή, παρά να επιβάλλουμε σε όλους τους χρήστες τα κατάντη στο τέλος για μέτρα πάρα πολύ επαχθή για την περιορισμό της μετάδοσης. Αυτό είναι ένα σημείο πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια λογική την οποία πρέπει να την ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ, Κορίνα Λεπάζ. Τελευταίος ομιλητής, ο Ρίχαρτ ε, Σίβερτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εξασφαλίσουμε ε, να υπάρχουν ασφαλή προϊόντα στην αγορά και εδώ έχει νομίζω ένα σημαντικό ρόλο να παίξει η Κομισιόν. Γιατί ξέρετε ότι σύμφωνα με τη συνθήκη έχουμε αυτή την αρχή της πρόληψης και θα πρέπει να εκτιμούνται έγκαιρα κινδύνοι που ενδεχομένω παρουσιάζονται στο μέλλον η Κομισιόν αναφέρεται πάντα στα επιστημονικά στοιχεία, αλλά υπάρχουν πολλές ε, αξιολογήσεις ε, που είναι ε, επιστημονικές και δεν είναι σύμφωνες με τις επιστημονικές αξιολογήσεις που αναφέρει η Κομισιόν. Δεν πρέπει εδώ να έχουμε έναν πίστης αλλά από την άλλη μεριά είναι καλό να εξετάζει κανένας πολύ προσεκτικά αυτά τα στοιχεία και νομίζω ότι η Κομισιόν και η ΕΦΣΑ παίζουν ένα μονομερή ρόλο. Το θέμα της ε, επιστημονικής βάσης και της ασφάλειας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να εξετάσετε και όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες ε, επιπτώσεις. Η Κομισιόν ε, έκανε μια πρόταση όσον αφορά την καλλιέργεια. Θα χαιρόμουν η Κομισιόν να μπορούσε να λύσει αυτό το μπλοκάσμα που υπάρχει στο Συμβούλιο για να μπορέσουν τα κρατημέλη να έχουν αυτή τη δυνατότητα γιατί ορισμένες χώρες, ορισμένοι ε, πολίτες είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το δεύτερο είναι επίσης σημαντικό. Η Κομισιόν θα πρέπει να φροντίσει να υπάρχει δυνατότητα επιλογής. Επιλογή σημαίνει ότι παραγωγή που θέλουν παραδείγματο χάρη να χρησιμοποιούν ε, ζωοτροφέ χωρί ε, γενικά τροποποιημένου οργανισμού να μπορούν να το κάνουν. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλάει κανένα για 100% καθαρότητα, αλλά αυτά τα κατόφλια δεν είναι επιστημονικά βασιζόμενα και αυτό είναι και η ε, παρατήρηση της Ρενάτε Ζόμερ που είπε ότι εν μέρη δεν υπάρχουν καν κατόφλια. Θα πρέπει λοιπόν να δράσει πάρα πολύ προσεκτικά η Κομισιόν όσον αφορά τους γενικά τροποποιημένους οργανισμούς γιατί μόνο αν είμαστε πολύ προσεκτικοί θα δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να κάνουν την επιλογή τους υπέρ ή κατά των προϊόντων αυτών. Και αυτό σχετίζεται βέβαια και με τη σήμανση των προϊόντων. Θα πρέπει οι πολίτες να ξέρουν ακριβώς τι τρώνε και όχι από την πίσω πόρτα ότι δεν μπορεί να το αποδείξουμε, είναι πολύ δύσκολο να το αποδείξουμε κλπ. Δεν είναι σωστό επιχείρημα σε μια τέτοια τεχνολογία που είναι τόσο σημαντική και που είναι πολύ δύσκολο να εκτιμήσουμε τις επιπτώσεις. Θα πρέπει η Κομισιόν να έχει κατά νου καλύτερα το μέλλον και να μην ε, ε, δρά μόνο προς συμφέρον μια συγκεκριμένη βιομηχανίας. Θα πρέπει, όπως σας είπα, να εξτάσουμε τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και εκτός αυτού είναι το θέμα και πολιτικό. Η Κομισιόν να μην έχει με τα λεγόμενα επιστημονικά επιχειρήματα κατά αυτόν τον τρόπο. Θα ήταν αυτό μοιραίο για όλο τον τομέα. Και γι' αυτό η Κομισιόν εδώ έχει ένα ειδικό ρόλο να παίξει και ελπίζω ότι οι σκέψεις θα κινηθούν προς την κτέφηση αυτή και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. το και Κύριε Πούλε, θέλετε να απαντήσετε ή όχι. Μερικά λεπτά. Thank you, very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, για την περιβαλλοντική εποπτεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στο θέμα αυτό και γι' αυτό ακριβώς σας είπα ότι συνεργαζόμαστε με τις επιχειρήσεις και τα κρατημέλη ώστε να βεβαιωθούμε ότι αυτή τη στιγμή λαμβάνεται έγκριση για ένα γενετικό στροποποιημένο οργανισμό, υπάρχει παρακολούθηση μετά από την θέση του στην εμπορία. Και γι' αυτό ακριβώς οργανώνουμε και μια διάσκεψη στο Μάρτιο ώστε να δούμε... Ε, κατά πόσον εφαρμόζεται αυτή η παρακολούθηση μετά από την ε, τοποθέτηση του εμπόριου ενός προϊόντων. Τώρα, η Ευρώπη έχει την πιο συμπαγή και την πιο διεξοδική αξιολόγηση σε περιβαλλοντικά θέματα και σε γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς στον κόσμο. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος στον κόσμο που να κάνει την ίδια αξιολόγηση που κάνουμε εμείς. Αυτό για να καθησυχάσω τους ευρωβουλευτές, η νομοθεσία μας θέτει τις βάσεις όχι για την εμπορία, αλλά ώστε να βεβαιωθούμε ότι οτιδήποτε τίθεται σε εμπορία δεν είναι επιζήμιο για τη δημόσια υγεία. Όσον αφορά το κατόφλι, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται για τις ζωοτροφές δεν είναι μέτρα για να εγκρίνουν την παρουσία μη εγκεκριμένων γενετικών στροποποιημένων οργανισμών. Θέλουμε να καθορίσουμε μία μέθοδο και δυνατότητα δειγματοληψίας ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι όλες οι αρχές ελέγχους χρησιμοποιούν την ε, ίδια μέθοδο για να καθορίσουν τη μηδενική παρουσία, διότι υπήρχε κάποια παρανόηση στην εφαρμογή των ε, μέτρων. Το τεχνικό μηδέν ε, για τα μη εγκεκριμένα ε, για τις μη εγκεκριμένες ζωοτροφές εξακολουθεί να ισχύει. Όσον αφορά τώρα αυτό που ανέφερε ο κύριος Φαντάλε, πράγματι συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη και έχει συσταθεί μια ομάδα η οποία ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της για να συζητήσει αυτή τη νέα τεχνική ελέγχου και ε, έχουμε ζητήσει και τη γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ και μόλις ολοκληρωθεί η έκθεση θα ξαναέρθουμε εδώ για να το συζητήσουμε μαζί σας. Ξέχασα να απαντήσω και στην κυρία Σόμερ. Για το κατόφλι για τους σπόρους, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι οι σπόροι πρέπει να μην είναι επομολυσμένοι με γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και εξακολουθούμε να αξιολογούμε αν χρειάζεται κατόφλι για να επιτρέπεται ε, κάποια παρουσία η οποία είναι αναπόφευκτη. Αυτό όμως είναι ακόμα υπομελέτη, επομένως δεν μπορούμε να σας παρουσιάσουμε πρόταση από αυτού. Για την καλλιέργεια. Καταρχάς να σας συγχαρώ γιατί χάρη στην κυρία Λεπάζ μπορέσαμε να έχουμε γνωμοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ήταν θετική γνωμοδότηση για την πρότασή μας. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να επιτρέπεται στα κράτη-μέλη να αποφασίζουν εάν θέλουν να καλλιεργούν ή να μην καλλιεργούν γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς για κοινωνικο-οικονομικούς λόγους, για χρήση γεών ή για αγρονομικούς παράγοντες. Η πρόταση αυτή τη στιγμή είναι ακόμα μπλοκαρισμένη σε επίπεδο Συμβουλίου. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εγκριθεί αυτή η πρόταση, διότι εμείς πιστεύουμε ότι είναι δίκαιο να επιτρέπεται στο κράτος μέλος να επιλέξει πώς θα χρησιμοποιείται το έδαφος τους βάσει των δικών τους ε, συνθήκων. Και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σας, ε, διότι έβλεπε μπροστά στο μέλλον και δέχτηκε θετικά την πρότασή μας. Η εφαρμογή αυτή τη νομοθεσία είναι κάτι το οποίο είναι συνεχώ εν εξελίξη. Συνεχώ εργαζόμαστε ώστε να έχουμε μια πιο συμπαγή και καλύτερη εφαρμογή. Και με τη βοήθειά σας βέβαια είμαστε διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε επιχείρημα θέλετε να εξετάσουμε και ελπίζω να συμφωνείτε κι εσείς μαζί μας ότι ήμασταν όσο το δυνατόν ανοιχτοί για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και κύριε Βουλή για τις πληροφορίες αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν νομίζω πάρα πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση και κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχιστεί και θα επαναληφθεί που στο μέλλον. Τώρα θα περάσουμε στο επόμενο θέμα, την πράσινη ζώνη στην Ευρώπη. 12.500 χιλιόμετρα πράσινη ζώνη δημιουργήθηκε από το δεδρούν παραπέτασμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό για, τις, ε, για την ε, βιοπικιλομορφία. Χαιρετίζω την κυρία Χαλφόμα και ε, τον κύριο Γκαλντέτσι. Έχουμε ένα βίντεο εκεί και είναι πολύ καλή ευκαιρία αυτή για την προστασία της φύσης. Μπορούμε να αρχίσουμε. How is it starting? Yeah? Okay. You ο Κάι Φρόμπελ θα σχολιάσει αυτά που βλέπουμε στην οθόνη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ, κύριε βουλευτέ, σα ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σα παρουσιάσω αυτή την πράσινη ζώνη Ευρώπη. Πρόκειται για μια, έναν άξονα ενωμένων βιοτόπων στην Ευρώπη, ένα από τα πιο ελκυστικά κατά τη γνώμη μας προγράμματα στον κόσμο. Για να δούμε. Το 1989 η οργάνωση προσέγγισης του περιβάλλοντος Bund στη Γερμανία ξεκίνησε αυτή την πράσινη ζώνη, δηλαδή η διατήρηση των βιοτόπων που είχαν δημιουργηθεί στο φρικτό αυτό γερμανο-γερμανικό σύνορο. Ε, Μια δράση που τη χάνει έντονε υποστήριξη ε, στη Γερμανία. Το 2002 ο Μικάιλ Γκορμπάτζοφ επισκέφτηκε αυτή την πράσινη ζώνη και παρουσία του ανθρώπου αυτού που συνέβαλε στην εξάρρυψη του δρού παραπετάσματος γεννήθηκε αυτή η ιδέα της πράσινης ζώνης Ευρώπη το 2004 έγινε η πρώτη ε, πανευρωπαϊκή διάσκεψη στην Πράχα 24 ε, χώρε συμμετέχουν, εκ των οποίων 15 κρατημένες τη Ευρωπαϊκή Ένωση, 3 υποψήφιε και 4 ενδεχόμενε υποψήφιε και 2 χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία και Νορβηγία. Η IUCN, διεθνή Οργάνωση Περιβαλλοντική Προστασία, είναι εκείνη που έχει υπό την προστασία στην ιδέα αυτή. Πρόκειται για 12.500 χιλιόμετρα ε, ζώνης ε, βιοτόπων. Εδώ βλέπετε μία ομάδα μη κυβερνικών οργανώσεων που υποστηρίζουν αυτή την ε, προσπάθεια. Γιατί συνεργάζονται τόσες πολλές οργανώσεις, γιατί είναι τόσο ελκυστική αυτή η ζώνη. Το ιδιαίτερο είναι ότι υπάρχει εκεί μία ένωση βιοτοπών, 39 εθνικά πάρκα, 2.200 ε, προσταγόμενες περιοχές επίσης κατά την ε, κατονομικούς αυτής της ζώνης. Γιατί όμως εκεί υπάρχουν όλες αυτές οι φυσικές περιοχές ε, και ελκυστικές επίσης ελκυστικά επίσης τοπία πολιτιστικά όπως εδώ Βουλγαρία, Σερβία ε, ήταν ακριβώς το σιδερό παραπέτασμα που χώριζε τους ανθρώπους επί δεκαετίας και άθελα βοήθησε τη φύση. Και δεν είναι τυχαίο, αλλά το αποτέλεσμα της πρόσφατης ευρωπαϊκής ιστορίας το ότι ακριβώς εκεί που ενώνονται το ΝΑΤΟ και η Ρωσίβουνα της Βαρσοβίας δημιουργήθηκε ένα σημαντικό στοιχείο φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά προστατευόμενα ε, ζώα στην ε, Δυτική Ευρώπη και στην Ανατολική Ευρώπη και βλέπετε την ε, ζώνη αυτή την πράσινη που συνενώνει αυτά τα απειλούμενα είδη. Επίσης όμως η πράσινη ζώνη αυτή είναι έχει χαρακτηριστικά στοιχεία από τις γεωγραφικές ζώνες της Ευρώπης και Τώρα που υπάρχει η αλλαγή του κλίματος, γίνονται οι αλλαγές από βορρά νότο και φαίνονται σε αυτή την πράσινη ζώνη. Έχετε εδώ πέρα κάποιες εικόνες. η λίμνη το άλλο από τα σύνορα της Φιλανδίας Ρωσίας, η πράσινη ζώνη στη Γερμανία ή το ποταμός Δράου στην Ουγγαρία είναι κάτι που θεωρείται πάρα πολύ αξιόλογο ακριβώς λόγω της Ένωσης της ε, Φυσικής Προτασίας και της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Υπάρχουν διάδρομοι Ένωσης ε, για τη φύση. Υπάρχει εδώ η ανάγκη να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ζωής και να μην ε, περιοριστούμε μονάχα στην τεχνική υποδομή. Αυτή η πράσινη ζώνη θα ήταν του ακρογωνίου λήθος ε, για μια, ε, <clears throat> για μια υποδομή φυσική της Ευρώπης, κάτι που υπάρχει ήδη, δεν, δεν ε, σχεδιάζεται τώρα. Εδώ βλέπετε ένα πολύχρωμο, πολύμορφο σημείο παρουσίαση των ανθρώπων τη Ευρώπη, ε, τη φύση τη Ευρώπη. Αυτό που δεν φαίνεται ίσω στην εικόνα είναι ο ενθουσιασμό των ανθρώπων αυτών από 24 χώρε τη Ευρώπη που συνεργάζονται σε μια πράσινη ζώνη που είναι πάρα πολύ ευρωπαϊκή, σε μια ιδέα που είναι πάρα πολύ ευρωπαϊκή με όλες τις πτυχές που παρουσιάζει και οι άνθρωποι που συνεργάζονται εδώ και 10 χρόνια σε αυτό πραγματοποιούν κάτι που χρειάζεται η προστασία της φύσης στην Ήπειρό μας. Δηλαδή με μεγάλα οράματα ενθαρρύνονται, οράματα που ξεπερνάνε τα στενά σύνορα κρατών, οράματα που μπορούν να ε, κάπου στις ανάγκες ε, βιοποικιομορφίας στην Ευρώπη. Απ' την άλλη μεριά όμως οράματα που προσφέρουν κάποια σύμβολα, κάποιες συμβολικές εικόνες αν μου επιτρέψετε να σας πω, η Ευρώπη δεν πρέπει να ορίζεται μόνο με μία ένωση στον τομέα της οικονομίας. Η Ευρώπη δεν χρειάζεται μόνο και εν ώψη της ευρωκρίσης ε, μόνο την οικονομία, χρειάζεται περισσότερα κοινά ευρωπαϊκά σύμβολα και όσον αφορά τον τομέα της φύσης και του πολιτισμού. Και γι' αυτό παρακαλούμε και ελπίζουμε να υπάρχει αναγνώριση και υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πράσινη ζώνη Ευρώπης που είναι το μεγαλύτερο παγκοσμίω σχέδιο για την ένωση της φύσης πέρα από εθνικά σύνορα. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτος, ευχαριστούμε τον δόκτωρο Καϊφόρος και την δόκτωρο Ριάννα Μπατέτσης. Μπορεί να έρθετε και εσείς εδώ. Πραγματικά αξιόλογο φυσικό φαινόμενο μια πράσινη ζώνη. Είχα πάει στην Σλοβενία, στη Λιθουανία, στη Δανία περνάει. Δεν ξέρω. Είναι γνωστό στη Σλοβενία. Αυτή η πράσινη ζώνη είναι γνωστή στη χώρα σας. Έχετε κάτι να μας πείτε από αυτού. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά ομολογώ ότι δεν το γνώριζα το σχέδιο αυτό. Δεν το είχα ποτέ ακούσει. Αλλά μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το γνώρισατε σήμερα. Η συνάδελφος είναι νέα στο κοινοβούλιο εδώ. Στην Λιθουανία το γνωρίζετε αυτό, γιατί υπάρχει εκεί αυτό το πράσινο κίνημα για την ελευθερία είναι και αυτό το τμήμα της ιδέας ίσως. E, Ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίασή σας. Θα ήθελα να υποστηρίξω τη συνάδελφο από τη Σλοβενία. Θεωρώ ότι το πρόγραμμα αυτό δεν είναι αρκετά γνωστό στο ευρύ Και Ελπίζω η παρουσίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας δώσει το ένασμα για να το συζητάμε ε, περισσότερο. Οι οργανώσεις που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα είναι γνωστές, είναι αρκετά δημοφιλείς, αλλά η δραστηριότητά τους στον τομέα αυτό δεν είναι αρκετά γνωστές. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τρομόπουλος. Ε, μπορώ να σας πω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το, ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ε, θα ήθελα απλώς να το θέσω εδώ στη συζήτηση, θα είναι γνωστό στον εισηγητή μας ότι ε, υπάρχει μια αντίστοιχη πρωτοβουλία που στηρίζουν με πολύ μεγάλη ένταση οι πράσινοι ε, και διαχειρίζεται ο κύριος Μίχαελ Κράμερ και αφορά τη δημιουργία ποδηλατόδρομων με, στο παλιό παραπέτασμα, ας πούμε το Iron Curtain ε, Trail, το οποίο και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε ως δραστηριότητα και μέχρι κάτω τα Βαλκάνια και την Ελλάδα. Ε, είναι στην ε, ίδια κατεύθυνση και λογική και αξιοποιεί τις υπάρχουσες ζώνες φυσικής κοινωνικής ε, βλάστησης οι οποίες μπορούν εύκολα να αποδεχθούν δραστηριότητες ε, όπως το ποδήλατο ή ε, να αποτελούν διέξοδο για τους πολίτες. Yeah. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Δεν ξέρω, γνωρίζετε την ιδέα αυτή. Ναι, ναι, ναι, ναι. Την ιδέα είναι με τον Μιχαήλ Κράμερ και το Σιδερό Παραπέτας να συνεργαζόμαστε πάρα πολύ ξεκίνησε γύρω από το Βερολίνο με το τείχο εκεί και ο Μίχαελ Κράμερ μετά συγκεντρώθηκε στο σίδερουν παραπέτασμα. Συνεργαζόμαστε στενά, ούτω ώστε έτσι να προωθήσουμε και τον ε, τουρισμό φύση. Υπάρχει στην συνεργασία. Μια ερώτηση από μένα, λέει ο Τι περιμένετε τώρα εσείς από το Κοινοβούλιο ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά. Κοιτάξτε, δεν ήταν τόσο γνωστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε συγκεκριμένους ε, τοποθεσίες είναι γνωστό βέβαια, αλλά χαίρομαι που υπάρχει συνένεση από τους βουλευτές και θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας υποστηρίξει όσον αφορά την ανάπτυξη αυτού του μοναδικού συστήματος των ενωμένων βιοτόπων μακρύτερο ε, του, του κόσμου. Δεν είναι κάτι που που οργανώνουμε αυτή τη στιγμή, που, που προγραμματίζουμε αυτή τη στιγμή, είναι κάτι που υπάρχει ήδη. Και θα θέλαμε πραγματικά μια υποστήριξη, ε, παραδείγματος χάρη ένα πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Ζώνη ή τουλάχιστον μια αναγνώριση ε, μέσω ενός ψηφίσματος ενδεχομένως που θα μπορούσε να γίνει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αναγνωρίσει ακριβώς αυτό το σχέδιο στην Γερμανία ε, ξεκίνησε το 89 ήδη και σε εθνικό επίπεδο προσπαθήσαμε να το προωθήσουμε και θα χαιρόμαστε λοιπόν με τον ίδιο τρόπο να το προωθήσουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόεδρος. Α, μάλιστα. κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες ε, συμμετέχουν επίσημα ή μόνο μη κυβερνητικε οργανώσει. Όχι, όχι, κράτη-μέλη συμμετέχουν. Στη μία παρουσίασε εκεί φάνηκε υπάρχουν τα λεγόμενα National Focal Points που είναι στην κυβέρνηση, στην τοπική αυτοδιοίκηση και μετά υπάρχει και ο συντονισμό των εθνικών μη κυβερνητικών οργανώσεων αλλά και οι ίδιες κυβερνήσει συμμετέχουν. Και τελευταία ερώτηση από μένα. Επαφή προς την Κομισιόν. Υπάρχει, υπάρχουν αντιδράσεις. Τι έχετε να πείτε από αυτού. Ε, κοιτάξτε, ε, περισσότερο από επαφέ. Ευτυχώς ε, και μάλιστα θα ήθελα να ευχαριστήσω γι' αυτό. Υπάρχουν προγράμματα live ή που λαμβάνουν χώρα ακριβώς στο, στην πράσινη ζώνη. Το Queen Net στην κεντρική Ευρώπη, παραδείγματο χάρη, ένα πρόγραμμα live είναι πρωτοβουλίε κάποιων ε, κρατών που ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που δεν υπάρχει είναι ρητή αναγνώριση και ενίσχυση όλη τη ιδέας. Από την Νορβηγία, Φιλανδία μέχρι κάτω στα Βαλκάνια μεμονωμένα, ναι, πολύ καλή, πολύ στενή συνεργασία, αλλά όχι στο σύνολο, με όλες τις 24 χώρες.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 έχετε ένα τμήμα που στο χάρτη φαίνεται σαν τμήμα της Λετωνίας. Ο χάρτης μάλλον συγγνώμη λέει ότι είναι η Λιθουανία, αλλά στο χαρτί που μας δώσατε λέει ότι είναι η Λετωνία. Θα ήθελα να διορθώσετε το λάθος, είναι, ανήκει αλλού η περιοχή. Α, μάλιστα. Ένα ιδιαίτερο στη γεωγραφία. Θα το λάβουμε υπόψη μας και αν υπάρχει σφάλμα θα το διορθώσουμε. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα το ξέραμε, αλλά Κάπου έγινε λάθο. λάθος. ωραία. Τώρα θα ήθελα να προτείνω να προτείνουμε στου συντονιστέ αύριο το πρωί να υποβάλει μια ερώτηση προ την Κομισιόν για το πώ θα μπορούσε να ενισχύσει την πρωτοβουλία Πράσινη Ζώνη Ευρώπη για να δώσει αυτή την αναγνώριση, την υποστήριξη και ανάλογα με το αποτέλεσμα αυτής της συνομιλίας το επόμενο στάδιο θα μπορούσε να ήταν ένα ψήφισμα. Αλλά σύμφωνα με αυτό που συζητήσουμε στην Επιτροπή μας θα αρχίσουμε με μια ερώτηση προς την Κομισιόν. Μετά θα έχουμε μια συζήτηση όπου πάλι θα μπορούσαμε να σας καλέσουμε να συμμετάσχετε. Εάν δεν υπάρχουν περαιτέρω ερωτήσεις, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας παρουσιάσετε αυτό το πρόγραμμα εδώ. Πολύ καλό ήταν, γιατί πραγματικά δεν είναι παντού γνωστό. Και μπορούμε να αναλάβουμε την πρωτοβουλία στο Κοινοβούλιο να το κάνουμε πιο γνωστό και πιο επιτυχές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, η συνεδρίαση για σήμερα. Αύριο στις 10 συνεχίζεται με τις συνεδρίες επιτροπής μας. Και στις 7 το βράδυ είπαμε έχουμε ένα κοκτέιλ στην αίθουσα Γεούντι Μενούχιν. Και είναι όλοι προσκεκλημένοι. Και ευχαριστώ τους διερμηνείς.